Ladies and gentlemen, please be seated. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Μπορούμε πια να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε διερμηνία στις γλώσσες των τακτικών μελών. Η συνεδρίασή μας ε, μεταδίδεται σε απευθύνση μετάδοση. Και ας ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερησίας διάταξης της ε, διήμερης συνάντησης σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί όπου θα ξεκινήσουμε στις 9 το πρωί στις 9 το πρωί αύριο για το δεύτερο μέρος της συνεδρίασης αν δεν υπάρχουν ε, παρατηρήσεις ε, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη Τα πρακτικά της τελευταίας συνάντησης της 14ης Ιουλίου έχουν διανεμηθεί. Προθεσμία είναι μέχρι το για να υποβάλετε επιφυλάξεις ή σχόλια είναι μέχρι το τέλος της συνάντησης της Επιτροπής ΕΝΤΕ. Διαφορετικά δεν υποβάλλεται τίποτα θεωρείται ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Πρώτο σημείο της ε, επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι ανακοινώσεις της Προέδρου. Ενημέρωση Α, συγγνώμη, ενημέρωση από την ε, αποστολή της Επιτροπής μας στη Μολδαβία που έλαβε χώρα 20 με 23 Ιουλίου Τριμελής ήταν η αποστολή και εγώ είχα την τιμή να προεδρεύσω. Πήγαμε στο Τσισινάου με τον κύριο Σντρογεύσκη και την κυρία Ίνες Αγιάλα Ήταν εξαιρετικά επικοδομητικό το ταξίδι αυτό, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πήγαμε στο Τσισινάου σε μια εποχή κάπως ιδιαίτερη διότι δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης. Μας υποδέχθηκαν ε, όλες οι σημαντικές ε, προσωπικότητες ε, της ε, πολιτικής σκηνής στη Μολδαβία. Αποφασίσαμε να κρατήσουμε χαμηλό προφίλ χωρίς μεγάλη παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης λόγω αυτής της ευαίσθητης από πολιτική άποψη εποχής. Φυσικά, κύριος σκοπός μας ήταν να αξιολογήσουμε τις προκλήσεις και τις επιδόσεις της αποστολής της Ευρωπαϊκής, ε, της Τεχνικής Αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συμβουλευτικής Αποστολής που προσέφερε αρρωγή στην Ουκρανία και τη Μολδαβία για τον έλεγχο των συνόρων. Σε μια κατάσταση αρκετά επισφαλή, εξαιρετικά δύσκολη, λόγω της προσάρτησης της Κρυμαίας τις δραστηριότητες ε, στην περιοχή της παγωμένης ε, ε, ένεξης στην υπερδυνιστερία θα έχετε λάβει όλοι σας την έκθεση από την αποστολή μας αλλά συμφωνούμε όλοι ότι η παρουσία της EUBAM εκτιμάται ιδιαίτερος και είναι αναγκαία σε μεγάλο βαθμό εκεί στην περιοχή. Δεν θέλω όμως να κάνω την ενημέρωση μόνη μου. Επιτρέψτε μου λοιπόν να δώσω το λόγο και στους ε, λοιπούς συμμετέχοντες. Να ζητήσω λοιπόν από τον κύριο Σδρογεύσκη πρώτα και μετά από την κυρία Αγιάλα να πάρουν τον λόγο για μια ενημέρωση προς τα μέλη της υποεπιτροπής ε, σε σχέση με τις δραστηριότητες της αντιπροσωπείας. Ε, κύριε Σδρογεύσκη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πιστεύω πως η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή. Και η Πρόεδρος ήδη ανέφερε τα σημαντικότερα στοιχεία της έκθεσης αυτής. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, είναι μια εξαιρετική έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ αυτό. Κυρία Γιάλα, θα θέλετε κι εσείς να συνεισφέρετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ αναγνωρίζω ότι κάνετε μία άψογη σύνοψη των εμπειριών μας, πολύ διδακτική, όπως είπατε και εσείς. Ήταν μια εποχή σχηματισμού ε, κυβερνητικού συνασπισμού Πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Γραμματεία και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτόπου, διότι μας βοήθησε πάρα πολύ στη διοργάνωση των επισκέψεων, ε, που ήταν ποικίλε, ε, είδαμε την κατάσταση από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Στην, ε, η Μολδαβία χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες ευαισθησίες, από μια πολυμορφία, ποικιλομορφία, το πανόραμα ήταν αρκετά περίπλοκο και ρευστό, πάντως η ελπίδα εκείνη την εποχή ήταν ότι θα σημαντιστεί ένας ε, ε, κυβερνητικός συνασπισμός ε, αποτελεσματικός και χωρίς συγκρούσεις. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η επίσκεψη, μας επέτρεψε να ε, εξετάσουμε την κατάσταση αυτή η οποία θα περιπλακεί πιστεύω τους επόμενους μήνες σε σχέση με την Ουκρανία και τη Ρωσία, τι θα γίνει με τους πρόσφυγες. Μας ε, ε, επέτρεψε να αποκτήσουμε μια πολύ καλή εικόνα των διαφόρων ευαισθησιών ε, που επικρατούν στην Μολδαβία. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να συμμετάσχω και ευχαριστούμε πολύ και για την προεδρία σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Αγιάλια. Σας ευχαριστώ όλους για την συνεργασία λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ και τη γραμματεία σχετικά με την ε, μόνιμη αντιπροσωπεία. Πιστεύω πως ε, η αντιπροσωπεία ήταν εξαιρετικά προετοιμασμένη σχετικά με όσα είχαν συμφωνηθεί. Μάλιστα ταξιδέψαμε σε μια πολύ δύσκολη χρονική στιγμή για την περιοχή αυτή. Πριν μεταβούμε εκεί είχαμε Έντονε διαβουλεύσεις. Προσπαθούσαμε να εξετάσουμε το πόσο συνετό είναι να πάμε εκεί, αν θα έπρεπε καλύτερα να αναβάλουμε το ταξίδι, όμως στο τέλος αποφασίσαμε να τηρήσουμε το πρόγραμμά μας και πιστεύω πως ήταν πολύ συνετή απόφαση. Η Δημοκρατία της Μολδαβίας αυτή την περίοδο περνάει δύσκολες ώρες. Όλοι βλέπουμε τι έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου με τις μαζικές διαδηλώσεις. Και αυτό είναι μια έκφραση μιας απογοήτευσης ή μιας ασάφειας, μιας έλλειψης σιγουριάς των πολιτών προς την κυβέρνησή τους. Και οι διαδηλώσεις το έδειξαν αυτό. Οι διαδηλώσεις ήταν υπέρ της Ευρώπης, υπέρ της Δύσης. Και όπως είπα διατυπώθηκε μια δυσπιστία για την κυβέρνηση της Μολδαβίας. Η οποία είχε να κάνει με τις ε, με την κατεύθυνση που έχει πάρει η κυβέρνηση. Ο λαός όμως έδειξε ότι είναι υπέρ της Ευρώπης. Κάτι που άλλωστε ήταν και δική μας εκτίμηση όταν πήγαμε εκεί. Αυτή τη στιγμή η Μολδαβία ανήκει σε μια ομάδα χωρών που παρουσιάζουν τις ε, μεγαλύτερες δυσκολίες. Είναι περίπλοκα τα πράγματα εκεί. Ο κόσμος αντιμετωπίζει δυσκολίες κάθε είδους και η κυβέρνηση δεν βοηθά ώστε να επιληθούν τα προβλήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο νέων εκλογών, κάτι που πιστεύω θα δώσει στους πολίτες ε, ένα αίσθημα ασφάλειας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, συμμετοχή σας στην αντιπροσωπή αυτή. Τώρα θα αρχίσουμε την ε, συζήτηση με τα υπόλοιπα μέλη που θα ήθελα να συζητήσουν το θέμα. Νομίζω πως μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Α, με συγχωρείτε. Η κυρία Γιάτεν Μάκη, έχετε το λόγο. Α, δεν συζητάμε ακόμα το σημείο για το εμπόριο όπλων. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θα περάσουμε ευθύ αμέσω σε αυτό το σημείο, στι εξαγωγέ όπλων. Ε, παρακαλώ. Θα μιλήσω σου ειδικά, οπότε παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αυτή την έκθεση και που μου τη συνέστησαν. Η Πρόεδρος ζητά από την ομιλήτρια να διακόψει για λίγο για να ανακοινώσει η Πρόεδρος τη διαδικασία αυτού του σημείου. Λοιπόν, περνάμε αμέσως στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. που είναι η πρώτη εξέταση ενός ε, σχεδίου έκθεσης ε, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων και την υλοποίηση της κοινή θέσης 2008-944. Η συγκητρία είναι η κυρία Μπόντιλ Βαλέρο και το σχέδιο έκθεσης υποβλήθηκε για μετάφραση τον Ιούνιο, αν έχω καταλάβει καλά. Και τώρα έχουμε την πρώτη εξέταση. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 23η Σεπτεμβρίου 2015, 12 το μεσημέρι. Στην αίθουσα βρίσκεται και ο κύριος Πιέρ Αρνό Λότον, της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου ε, ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και θα ακούσουμε και τα δικές του παρατηρήσεις κατά τη συζήτηση σε σχέση με το σχέδιο έκθεσης. Μετά από τη συζήτηση όμως θα θέλαμε να γίνει και μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο ε, για να δούμε ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το καθεστώς ελέγχου της εξαγωγής όπλων. Κυρία Βαλέρο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξαναρχίσω, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ όλες και όλους που μου ανέθεσαν και μου εμπιστεύτηκαν αυτή την έκθεση. Για τρία χρόνια ε, μελετούσα το θέμα των συστημάτων ελέγχου εξαγωγών όπλων ε, και στην ε, Σουηδία η πίεση της, από την κοινή γνώμη και από τις οργανώσεις των πολιτών ήταν πολύ ισχυρή έτσι ώστε να σταματήσουμε να, συνεχίσουμε, να μην συνεχίσουμε πια να εξάγουμε όπλα σε καταπιστικά καθεστώτα όπως η Σουηδική Αραβία. Ε, τα όπλα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την άμυνα των χωρών μας αλλά οι τα όπλα που εξάγουμε δεν θα πρέπει να καταλήγουν στα χέρια ανθρώπων και οργανώσεων που μπορεί να αποτελέσουν απειλή ε, για την ασφάλεια άλλων ή και τη δική μας. Για αρκετά, για πολλά χρόνια έχουμε δει τέτοιου είδους απειλές εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και η βιομηχανία, ο κλάδος ε, προσπαθεί να βρει συνεχώς καινούργιες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να αυξήσει εξαγωγές. Θα πρέπει όμως να βλέπουμε τα πράγματα πιο μακροπρόθεσμα. Μια συμφωνία που ξεκινάει σήμερα μπορεί να ολοκληρωθεί μετά από πολλά χρόνια με πολλές ε, παραδόσεις όπλων ε, στο ενδιάμεσο. Θα πρέπει λοιπόν αυτές οι πωλήσει, αυτές οι εξαγωγές να γίνονται με πολύ συγκεκριμένους και αυστηρούς όρους. Τώρα έχουμε τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική για παράδειγμα. Εκεί έχουμε μακροπρόθεσμα, μακροπρόθεσμες συμβάσεις εδώ για πολλά χρόνια. Έχουμε προσπαθήσει να πουλήσουμε όπλα σε αυτές τις χώρες ε, για πολύ καιρό. Τώρα όμως γνωρίζουμε τι προβλήματα υπάρχουν. Τα όπλα καταλήγουν πολλές φορές στα λάθος χέρια και έχουμε χάσει σε ένα μεγάλο βαθμό τον έλεγχο. Σε ό,τι διαφορά τα ελαφρά όπλα, η έκθεση Europa για τις εξαγωγές τους ε, ανέφερε ότι αυτά επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα χέρια οργαν... Ε, κλιματικών οργανώσεων και τρομοκρατικών οργανώσεων. Επίση, πουλάμε πολλά όπλα στη Ρωσία που επίση μπορεί να αποτελέσει απειλή. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί με τα συστήματα ελέγχου των εξαγωγών και να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια κοινή θέση. Ε, αντί απλώ να ηθικολογούμε, ε, προσπάθησα να εστιάσω την έκθεσή μου σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα στα οποία πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να παίξει ρόλο, και ώστε να βελτιωθούν οι κανόνε ή η συμμόρφωση με του κανόνε. Ε, περιμένω τις ε, τροπολογίες σας ε, και θα τις συζητήσουμε με τους κοιόδης ηγητές αργότερα δεδομένου ότι ενδεχομένως δεν θα έχουμε χρόνο να τα δούμε όλα σήμερα. Να δω τρία πράγματα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, την, την αλλαγή της κατάστασης ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές πωλήσει μας πηγαίνουν σε γειτονικέ χώρες ε, προβληματικές χώρες και η, η βιομηχανία όπλων θα πρέπει να αναρωτηθεί ε, και εμείς όλοι μαζί γιατί κατασκευάζουμε όπλα και πώς θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Ε, δεν θέλουμε να γίνονται πωλήσει που θα μειώσουν τη δική μας ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να ακολουθούμε συγκεκριμένους κανόνες όπως η συνθήκη εμπορίας όπλων, ε, η κοινή θέση και το εγχειρίδιο χρήστη. το εγχειρίδιο χρήστη για παράδειγμα θα πρέπει ε, να ε, τηρείται κατά γράμμα και θα πρέπει να πάρουμε πολύ στα σοβαρά το θέμα των εξαγωνόπλων διότι αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να ξαναδούμε τους κανόνες μας και δεν θα πρέπει να περιμένουμε τόσο όσο παλιότερα για να ε, ε, εκδίδουμε εκθέσεις. Η βασική ιδέα είναι ότι δεν θα πρέπει να πολλούμε όπλα σε χώρες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα όπλα για να καταπιέσουν τους πολίτες τους. Μπορεί κανείς να πουλήσει ένα υποβρύχιο με τον ίδιο τρόπο που πουλάει εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών στην αστυνομία. Στην αστυνομία, στην Σουηδία έχουμε εθνικές κατευθυντήρες γραμμές ε, εξετάσαμε πολύ καλά την κατάσταση στη χώρα μας ε, σε περιπτώσεις παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν χορηγούμε ή αναστέλουμε άδειες, εξαγωγικές άδειες όπλων. Θα πρέπει κανείς να είναι πολύ αυστηρός από την άλλη μεριά όμως δεν θα πρέπει να παρεμποδίσουμε το έργο χωρών που έχουν ακόμα πιο αυστηρές, αυστηρούς κανόνες από ότι εμείς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υπάρχουν ε, χώρες οι οποίες έχουν πάει πιο μακριά. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο κοινό παρανομαστή, αλλά ορισμένε χώρες θα μπορούν να πάνε ακόμα πιο μακριά. Το ένα άλλο θέμα είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία. Ε, ως ευρωβουλευτές και ως βουλευτές, εθνικοί βουλευτές, πρέπει να ελέγχουμε τις κυβερνήσεις μας. Αλλά σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι μας. Θα πρέπει όλοι να κάνουν το ίδιο. Και το κοινό και οι βουλευτές θα πρέπει να μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις σέβονται τους κανόνες. Και οι εκθέσεις για αυτά τα θέματα θα πρέπει ε, να είναι και έγκαιρες και επίκαιρες και πιο προσβάσιμες. Ε, και στον ορισμένο μένω Αθηνών το θέμα των <clears throat> εξαγωνόπλων και είμαι σίγουρη ότι η ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, υπερτερούν έναντι των εξαγών για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Uh, thank you, Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαλέρο. Τώρα το λόγο θα πάρουν οι σκιώδεις συζητητές. Αυτό μας ε, έχει δώσει κάποιες δυσκολίες διότι υπάρχουν απόντες και δεν έχουν ειδοποιήσει όλη τη γραμματεία. Αλλά το ΕΛΚΑ σίγουρα έχει ειδοποιήσει. Κύριε Κέλαμ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν αναγκαία αυτή η έκθεση για αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Για πολλά χρόνια παρατηρεί το κατάχρηση των εξαγωγών όπλων με παρεκτροπή των όπλων από μια χώρα σε άλλη. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να εκτιμήσουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια κατά κάποιο τρόπο μοναδική θέση έχοντας εισαγεί το δικό της ε, σύστημα ελέγχου των όπλων όπως εκφράζεται στην κοινή θέση του Συμβουλίου για να πω και κάτι θετικό ε, να αναφερθώ στην παράγραφο 12 της έκθεσης όπου αναφέρεται η αναθεώρηση της κοινή θέση ε, της ΚΟΑΡΜΣ και τα συμπεράσματα που εξυπηρετούν τους στόχους του Συμβουλίου βρίσκεται, αυτό ευθυγραμμίζεται με την ε, συνθήκη ε, για τα όπλα. Είναι θετικό λοιπόν, ε, θετική ένδειξη. Φυσικά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτή η κοινή θέση που διατυπώνεται με αρκετά αυστηρούς όρους και επιτρέπει ε, και ακόμη πιο αυστηρή προσέγγιση ε, και εφαρμογή από τα επιμέρους κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμοστεί πιο ομοιόμορφα. Υπό αυτή την έννοια καλωσορίζουμε τις online πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών, τις βελτιωμένες μεθόδους διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών και φυσικά ιδιαίτερα όσον αφορά την απόρριψη αδειών ε, για εξαγωγή όπλων από ορισμένα κράτη-μέλη, ε, είναι σαφές ότι οι πληροφορίε αυτές πρέπει να ανταλλάσσονται άμεσα μεταξύ όλων των κρατών μελών. Όπως ήδη ανέφερα, και αυτό είναι ένα σημείο που περιλαμβάνεται στην κοινή μας ε, θέση, υπάρχει ένας κίνδυνος παρεκτροπής των όπλων από την ε, χώρα παραλήπτη και να επανεξεχθούν. Εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Ταυτόχρονα εγώ ανησυχώ όσον αφορά τη σημερινή στάση προς αυτή την κατάσταση. Θα επιθυμούσα καλύτερη ενημέρωση για την Ευρωπόλ, όπως αναφέρεται στην παραγραφό 6, όσον αφορά την επανεισαγωγή πυροβολών όπλων από χώρε ε, στις οποίες έχουμε εξαγεί όπλα πίσω στην Ευρώπη. Όπως αναφέρεται είναι ένα σενάριο, αλλά όπως φαίνεται τα στοιχεία της Ευρωπόλ δεν επιβεβαιώνουν τέτοιες κινήσεις ρητά. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ε, και την ευρύτερη εικόνα της κατάστασης διότι ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ε, αναγνωρίζει ρητά το επιμέρους ε, δικαίωμα αυτοάμυνας και η αυτοάμυνα απαιτεί όπλα σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε γενικές λοιπόν γραμμές δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι τα όπλα είναι καλά ή κακά. Είναι καλά ή κακά ανάλογα με τους χρήστες τους. Και φυσικά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους χρήστες. Ε, όπως περιπτώσεις καλής χρήσης ως, αποτρεπτικούς, ως αποτρεπτικό παραγόντων, αλλά φυσικά ε, υπάρχουν Περιπτώσει όπου η ισορροπία αυτή μεταξύ αποτροπής και χρήση χρήσης ε, είναι έθραυστη. Α δούμε την κατάσταση μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν έχει όπλα ούτε για να υπερασπιστεί τον εαυτό τη και πολλά κράτη-μέλη αποφάσισαν να εξαγούν αμυντικά όπλα στην Ουκρανία. Τέτοιε περιπτώσει επίση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Και σε ορισμένε άλλε περιπτώσει τα όπλα χρησιμεύουν για την επιδευτική σταθερότητα όπως σε ορισμένες περιοχές του Ιράκ και της Συρίας όπου τα όπλα που δόθηκαν στους Πεσμεργά οι οποίοι μάχονται κατά του Ισλαμικού κράτους στους ε, Γιαζίδη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι κατανοητό η αναγκαιότητα ύπαρξη των όπλων οπότε γενικά έχω να πω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να παρέχουμε μια προσέγγιση σταθερή ε, ε, εξισορρόψης ε, σε αυτό το πολύ το θέμα. Και αν χρειαστεί θα χρειαστεί να ορίσουμε πιο αυστηρούς όρους για τις εξαγωγές όπλων. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τις γενικότερες πτυχές της όλης κατάστασης Επίση, ε, θα υποβάλουμε τροπολογίες οι οποίες ελπίζω να συμβάλλουν ε, στην βελτίωση και στην επίτευξη καλύτερη ισορροπίας για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλεμ. Για τους Σοσιαλδημοκράτε, η κυρία Ένα Σαγιάλια, σκιωδή συγγετρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν σας ε, στείλαμε πιο νωρίς το όνομά μου, αλλά πράγματι είμαι σκιώση ηγητρία στην έκθεση της κυρίας Βαλέρο. Την ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και για αρκετές από τις προτάσεις της. Να κάνω τα εξή ε, σχόλια. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, το είπαμε και πριν. Θα ήθελα ήδη στον τίτλο να μην μιλάμε μόνο για εξαγωγές, αλλά όχι μόνο για έλεγχο των εξαγωγών, αλλά ε, συγγνώμη, όχι μόνο για εξαγωγές, αλλά και για έλεγχο εξαγωγών, γιατί αυτή είναι η λειτουργία την οποία προσπαθούμε να ρυθμίσουμε. Τα οκτώ κριτήρια της κοινή θέση υιοθετήθηκαν ε, κατά τη διάρκεια της Ισπανική ε, Προεδρίας, οπότε ε, κατά κάποιο τρόπο αισθανόμαστε και πιο εμπλεκόμενοι με την κοινή θέση ω Ισπανοί. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω για τη δουλειά της και να τη ρωτήσω κάποια πράγματα. κάνει λόγο για σειράξεις ή συγκρούσεις. Φαντάζομαι ότι εννοεί πως είναι σημαντικό ε, να περιορίσουμε τα επιθετικά όπλα. Όμως ορισμένες ε, περιπτώσεις όπως για παράδειγμα στην ε, Ουκρανία ή και στη Σύρια ε, έχουμε ε, κάποιον επιτιθέμενο και κάποιον αμυνόμενο που πολλές φορές η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί να τον ε, βοηθήσει ε, χάρη στην υποτιθέμενη εφαρμογή της ουδετερότητας, της αρχής ουδετερότητας. Και εμείς στην Ισπανία είχαμε μια παρόμοια κατάσταση. κάποια στιγμή έπρεπε να ανοίξουμε τα στρατόπεδα, να ανοίξουμε τις αποθήκες και να δώσουμε όπλα στον κόσμο για να αμυνθεί εναντί μιας επιθεση ε, που δεχόταν. Ε, οπότε ε, καμιά φορά χρειάζεται για τη δική μας άμυνα να κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους αμυνόμενους. Μετά, γίνεται λόγος επανειλημμένος στην έκθεση για την Αραβική Άνοιξη, κάτι που μου δημιουργεί μια σύγχυση. Για, μέρα, για μένα η ε, Αραβική Άνοιξη ε, είναι, ήταν κάτι θετικό, διότι οδήγησε κάποιες αλλαγές. Τώρα, από εκεί πέρα, άλλο θέμα είναι οι επιπτώσεις και το πώς τη διαχειριστήκαμε. Όμως, ε, τα διδάγματα της ε, Αραβικής Άνοιξης δεν είναι μόνο αρνητικά. Θα πρέπει να γίνει σαφές για το τι μιλάμε, για, το, για ποιο πράγμα μιλάμε όταν αναφερόμαστε στην Αραβική Άνοιξη. Μετά, έχουμε, ε, έχει καθυστέρησε πάρα πολύ η ετήσια έκθεση και συμφωνώ. Ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από σημαντική έλλειψη συγκρίσιμων στοιχείων. Πολλές χώρες δεν έκαναν τα καθηκοντά τους, δεν έκαναν τη δουλειά που έπρεπε. Εμείς ε, στην, έκθεση, στην Επιτροπή Μεταφορών τα καταφέραμε και κάναμε καταλόγους ε, με μαύρους καταλόγους ας πούμε με χώρες τις οποίες ε, ε, επιτρέπεται και, που απαγορεύεται και άλλους καταλόγους με χώρες ή με επιχειρήσεις τις οποίες επιτρέπεται να δίδονται άδειες. Το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και εδώ δηλαδή καταλόγους θετικούς και αρνητικούς με επιχειρήσεις οι οποίες ε, απαγορεύεται ή επιτρέπεται να διδόνται εξαγωγικές άδειε. Επίσης μιλήσατε και για κυνηγητικά και όπλα και για όπλα σκοποβολής. Ε, πράγματι στην συνθήκη ε, ε, εμπορίου όπλων υπάρχει ειδικό καθεστώς για αυτά τα όπλα και θα έπρεπε να τα δούμε πράγματι ένα κινητικό όπλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ένα πόλεμο αλλά η, ε, η κανονική του χρήση είναι κάποια διαφορετική ε, οπότε ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να τα δούμε όλα τα όπλα με τον ίδιο τρόπο ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια διάκριση για τα κινητικά όπλα ή και για τα όπλα που χρησιμοποιούνται στη σκοποβολή Επίσης λέτε ότι χρειάζεται να εντοπίσουμε και άλλες ε, χρήσεις ε, τεχνολογιών όπως για παράδειγμα τα μη επανδρομένα αεροπλάνα, αεροσκάφη ε, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και προϊόντα ρομποτικής που έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Νομίζω, οι ειδικοί μας λένε ότι είναι σημαντικό να δούμε πως η χρήση αμυντική επιθετική όπλων και τεχνολογίας ε, ε, να συμπεριθεί και αυτή για να καλυφθεί. Επίσης για το λαθρεμπόριο όπλων. Ε, έχω να πω το εξή Ορισμένα όπλα κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξάγονται και μετά επανισάγονται Το λέτε και εσείς στην έκθεσή σας όλη αυτή, όλο αυτό το εμπόριο, όλη αυτή η διακίνηση όπλων που δημιουργεί και τρομακτικά κέρδη θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο κείμενο να προσθεθεί, να υποβάλουμε κάποια τροπολογία ενδεχομένω. θα υποβάλουμε εμείς σε τροπολογία σε ό,τι αφορά αυτή τη διακίνηση όπλων και την οικονομική της διαχείριση ε, τα κέρδη τα οποία μπορούν να προκύψουν ε, από την καταπολέμηση τέτοιου είδους παράνομου διακίνησης. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κασοντανισκή από την ομάδα ECR. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να τοποθετηθώ για την έκθεση αυτή. Φυσικά στηρίζω την ε, κατεύθυνση της συζητήτριας. Έχω κάποιες παρατηρήσεις βέβαια για τα σημεία C και D των αιτιολογικών σκέψεων. Αναφερθήκατε σε αυτά εδώ κατονομάζεται η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως εξαγωγής όπλων και αναφέρεται και ο ρόλος τους ως εξαγωγής. Φυσικά τα σημεία αυτά αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό να αναφερθούμε συγκεκριμένα σε ορισμένα κράτη. Επίσης, το σημείο 21 σχετικά με τη διαφάνεια, όπου παρατηρείται με λύπη ότι μόνο 21 κράτη-μέλη υπέβαλαν πλήρη συμμετοχή στην 16η εκτήσια έκθεση. Αναφέρεται ότι η Γερμανία δεν παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τις πραγματικές εξαγωγές. Η Γερμανία είναι μία από τις χώρες που εξάγουν σε μεγάλο αριθμό οπλικά συστήματα, νομίζω είναι τρίτη. Και αυτό είναι ένα εθνικό θέμα, δεν αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, έχω και μία ερώτηση. Αναφερθήκατε στις ευθύνε των κρατών ε, μελών ε, και επίσης λείπει από την έκθεση μια αναφορά στις εξαγωγές όπλων προς τη Ρωσία, για παράδειγμα μετά την εισβολή στη Γεωργία. Και πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό. Ότι δηλαδή ο ρωσικός στρατός προχώρησε λίγα χιλιόμετρα πιο κοντά στην Γεωργία και ανέβηκε φυσικά το επίπεδο ανασφάλειας στην χώρα. Πώς ε, λοιπόν θα μπορέσουμε να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά σε αυτά τα κριτήρια. Ιδιαίτερα όταν στην περίπτωση της Ρωσίας δεν τηρούνται αυτά τα κριτήρια, αυτές οι προϋποθέσεις. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Η Rheinmetall για παράδειγμα, γερμανική εταιρεία, η οποία δημιούργησε ένα κέντρο κατάρτισης στη Ρωσία και δαπανήθηκαν πόροι για αυτό το κέντρο. Και επίσης, όσον αφορά την ε, παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας, νομίζω πως και αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην έκθεση, έτσι ώστε να αποκομίσουμε μια πληρέστερη εικόνα σχετικά με, την εξαγωγή, με τις εξαγωγές όπλων και τη σχετική ε, τεχνολογίας για διπλό σκοπό. Χρειάζεται λοιπόν να αναφερθεί η Ρωσία. Τώρα περνάμε στις αραβικές χώρες, στη Μέση Ανατολή, στην Αγγής Ανατολή, στις χώρες νότιας γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Και φαίνεται πως η Ρωσία θα γίνει και αυτή ένα σύμμαχος στον αγώνα κατά του Ισλαμικού κράτους. Χρειάζεται λοιπόν να συμπεριληφθούν και αυτές οι αναφορές στην έκθεση έτσι ώστε να είναι πληρέστερη. Επίσης και ο ρόλος του Ασάντ στις εξαγωγές όπλων. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία, Η του Άλντε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Βαλέρο για την πολύ σημαντική αυτή έκθεση. Έχετε κάνει εξαιρετική δουλειά και όπως υπόθηκε το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Θα περάσω στα αγγλικά λέει η ομιλήτρια. Για πολλά χρόνια ζητούσα αύξηση της διαφάνειας των εμποριόπλων και η κοινή θέση και η διεθνή συνθήκη για τον πορεοπλόν είναι βήματα προς σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, το πρόβλημα φαίνεται να είναι ότι η εφαρμογή της διαφάνειας και των ρητρών υποβολησάν εκθέσεων. Οπότε πρέπει να πω ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την κυρία Βαλέρο. Πρέπει να υπάρξει κάποια τυποποίηση των εκθέσεων με προθεσμίες υποβολής των ε, στοιχείων ε, αδειοδότησης και εξαγωγών. Βέβαια βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της ε, έγκρισης της συνθήκης από την Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε τέθηκε σε ισχύ τέλη του περασμένου έτους. Οπότε στην αρχή βέβαια της εφαρμογής μιας τέτοιας συνθήκης πάντα υπάρχουν δυσκολίες αλλά να υπενθυμίσω τα κράτη-μέλη ότι τα ίδια έχουν συμφωνήσει επί των οκτώ κριτηρίων της κοινή θέση και οι κυβερνήσεις και τα κράτη-μέλη πρέπει να ε, εκπληρώσουν την υποσχέσή τους. Και πάντα αυτό είναι το πρόβλημα ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι κυβερνήσεις ε, κάνουν διάφορες υποσχέσεις τις οποίες δεν τηρούν. Ε, κάτι άλλο τώρα. Πρέπει να πω ότι διαφωνώ λίγο για τη στάση της κυρία ε, Σβαλέρο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εξοπλιστική Βιομηχανία. Διότι από όσο καταλαβαίνω ότι οι δημοσιονομικές περικοπές ε, οδηγούν τις εταιρείες της Ευρώπης να αναζητήσουν αγορές αλλού. Αυτή είναι η λογική των επιχειρήσεων και είναι απόλυτα κατανοητή. Όμως ρόλος των κυβερνήσεων είναι όλο αυτό να λαμβάνει χώρα ε, τηρώντας την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η θέση του Άλντε. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστούμε, ο κύριο Στέτινα. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Και εκεί θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, ό,τι φορέστε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα να πω ότι ο φιλιρινισμός μπορεί να είναι και επιζήμιος μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Θυμηθείτε τι έγινε με την Jane Φόντα που διαδήλωνε κατά του πολέμου στο Βιετνάμ. Σίγουρα είχε καλές προθέσεις, όμως στο τέλος όλα αυτά οδήγησαν στη, στην διάσπαση της χώρας και στο μισό της χώρας κάτω από τον κομμουνιστικό ζυγό. Το θέμα είναι εδώ για μένα σε ποιον πηγαίνουν τα όπλα. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της Συρία και της Ουκρανίας. Η Ουκρανία χρειάζεται όπλα έτσι ώστε να μπορεί να αμυνθεί. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε ήδη. Ωστόσο πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την αναφορά, ιδιαίτερα μάλιστα αναφερόμενοι και στις χώρες ε, οι οποίες βοηθούν την Ουκρανία. Η δική μου χώρα πριν από μερικά χρόνια είχε στείλει πυρομαχικά στο Κουρδιστάν στο Ερμπέλ, την πρωτεύουσα του ε, Κουρδιστάν στο Ιράκ. Είχε στείλει λοιπόν 500 τόνους πυρομαχικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν από την πολεμική αεροπορία. Ζήτησα από τον αρμόδιο Υπουργό, Υπουργό Άμυνας της χώρας μου περισσότερες πληροφορίες και κατόπιν έμαθα ότι είχαν σταλεί όπλα και στο κομπάνι εκτός από το Έρμπιλ όπου οι Κούρδοι της Συρίας πολεμούν το Ισλαμικό κράτος. Αυτές είναι εξαγωγές ε, όπλων οι οποίες είναι αναγκαίες. Γι' αυτό θα ήθελα να το υποβάλω ως τροπολογία και θα ήθελα να συμμετέχω στην ε, κατάρτιση της έκθεσης. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γκόμες. Χαίρομαι που τελικά το Κοινοβούλιο για μια ακόμα φορά ασκεί τα δικαιώματα ελέγχου που έχει. Το Κοινοβούλιο έχει να παίξει αποφασιστικό ρόλο γιατί για πολλά χρόνια ακόμα και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπήρχαν τρομακτικές αντιστάσεις έτσι ώστε η κοινή θέση να γίνει δεσμευτική μεταξύ των κρατών μελών. Και δεν είναι τυχαίο. Παρόλο ότι υφίστατο ήδη ένας ε, ε, κώδικα συμπεριφοράς, μη δεσμευτικός βέβαια, ε, ε, δεν, ε, δεν τον τηρούσαν πολλές χώρες και αντιδρούσαν έτσι ώστε στο η κοινή θέση να καταστεί δεσμευτική. Όμως κατέστη δεσμευτική επί Γαλλικής Προεδρίας το 2008 και το σύστημα ξαφνικά έπεσε ε, σε κενό διότι δεν υπήρχε κανένα όργανο ελέγχου ούτε καν το κοινοβούλιο. Οπότε η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη από ό,τι πριν. Η δική μου χώρα θυμάμαι, που δεν είναι η χειρότερη από όλες, είχε ένα σύστημα το οποίο ε, κοινοποιήθηκε, δηλαδή κοινοποιούσαμε τις εξαγωγές για αυτό το σύστημα εξαγών, αλλά υπήρχε και άλλο ένα σύστημα εξαγών από την αστυνομία και όχι από το στρατό, το οποίο δεν το Και είμαι σίγουρη ότι η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί και είμαι επίσης σίγουρη ότι δεν είναι η δική μου χώρα η μόνη ε, να το πω έτσι. Το είπε η κυρία Αγιάλα Σέντερ, το θέμα των, της εξαγωγής ε, των όπλων ε, κυνηγητικών ή αθλητικών όπλων, το οποίο πολλές φορές κρύβει τέτοιου είδους καταστάσεις διπροσωπείας. Κυρία Βαλέρα, η αθλητικων οπλων το οποιο πολλες φορες κρυβει τετοιου ειδους καταστασεις διπροσωπειας κυρια βαλερα έκθεσή σας είναι πολύ καλή. Θα πρέπει όμως να, μιλάμε, να μιλήσουμε λίγο και για το λόγο των ενδιάμεσων. Ε, υπάρχουν πολλοί ενδιάμεσοι ε, έμποροι όπλων. Ε, και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς. Άκουσα ότι αυτοί που επιτέθηκαν στο Σαγλίεμπτο αγόρασαν τα Καλάσνικοφ που χρησιμοποίησαν στην Κάρδη Μιντή στις Βρυξέλλες. Τα όπλα ήταν ε, κατασκευασμένα στην Ευρώπη και ήρθαν μέσω της Λιβύης. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την ε, εξαγωγή και επανεισαγωγή, ε, αυτό τον κύκλο που κάνει η διακίνηση των όπλων και αυτά επιστρέφουν στην πηγή τους. Επίσης έχουμε και τα εκρηκτικά ε, μικρές διατάξεις ή μηχανισμούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε τρομοκρατικές και άλλες δράσεις στη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως ε, κάποια στιγμή θα έρθουν και στην Ευρώπη και είναι ε, τρομακτικό το πώς τα κράτη-μέλη αγνοούν την κοινή θέση και την Συμφωνία Εμπορίου Όπλων μεταξύ άλλων. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε την ε, ε στήριξη της ΣΥΠΡΗ έτσι ώστε στην έκθεση αυτή να βάλουμε όσα στοιχεία μπορούμε για τις μη κοινοποιούμενες εξαγωγές των κρατών μελών. Για παράδειγμα γίνεται λόγος για την Ελλάδα, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Ε, τα, τις αναφέρει το κείμενο. Ε, την το πριν από 15 μέρες ήμουν στο Ιράκ, στην Ερμπίλ. Και εκεί μπορώ να συμφωνήσω. Ε, ε, ήταν χρήσιμη και είναι χρήσιμη η προμήθεια όπλων εκεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να γίνει με συντονισμένο τρόπο από τα κράτη-μέλη. Όχι έτσι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Στην Ερμπίλ οι άνθρωποι είναι πολύ χαρούμενοι με, το, με τα ε, αντιαρματικά μιλάν που τους έδωσε η Γερμανία ε, αλλά χρειάζονται πολύ περισσότερο εξοπλισμό για να πολεμήσουν τον Ισλαμικό στρατό ε, και ε, δεν τους το πουλάνε οι Ευρωπαίοι όχι για κανένα λόγο αλλά επειδή δεν συντονίζονται μεταξύ τους και με αυτόν τον τρόπο προδίδουν όλους τους Ευρωπαίους πολίτες όχι μόνο τους ανθρώπους του Ιράκ η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική και πρέπει να την ενισχύσουμε ε, προσθέτοντας όσο πιο συγκεκριμένα στοιχεία γίνεται έτσι ώστε να κατονομάσουμε τους κακούς μαθητές. Όταν αυτοί δεν συμμορφώνονται με τις ε, δεσμευτικές ε, υποχρεώσεις τις οποίες έχουν προσυπογράψει. Ευχαριστώ κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται πιστεύω να επαναλάβω πτυχές ε, στις οποίες συμφωνούμε, για παράδειγμα ε, για την κοινή θέση, για την ανάγκη ύπαρξης μιας ε, κοινή θέση, για τη συνθήκη, για το εμπόριο όπλων. Φυσικά αυτά είναι θέματα που τα καλώ ορίζω. Θα ήθελα να πω ότι στην, στις τελευταίες εξελίξεις της πολιτικής ασφαλείας βλέπουμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία μετά από την αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης έχουν ε, οπισθοχωρήσει, έχουν αλλάξει άποψη. Ορισμένες φορές αυτό συμβαίνει με τη δική του θέληση, όμως όποιες άλλες φορές ε, συμβαίνει μετά από την πίεση της κοινή γνώμης. Για παράδειγμα η στάση της ε, Γαλλίας με τους δύο Μιστρεάλ που δεν τους παρέδωσε τελικά στη Ρωσία. Επίσης αυτό το κέντρο άσκησης, κατάρτισης που συγκροτεί η Ράιν Μετάλλη στην Ρωσία. Αυτό το κέντρο αυτή τη στιγμή έχει αναστείλει προσωρινά την λειτουργία του φυσικά και Είμαι στη διάθεσή σα για περισσότερε πληροφορίε θα το ψάξω και εγώ ίδιο, διότι δεν θέλω να έχουμε τις λάθο εντυπωσει. Αυτά από τη μία. Από την άλλη, τα κράτη-μέλη φυσικά και χρειάζεται να έχουν μια κοινή θέση, όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται και μια κάποια εναρμόνιση τη εφαρμογή όλων αυτών των κανόνων διότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, υφιστάμενες οδομές οι οποίες χρειάζονται αρμόνιση. Επίσης από την άλλη σκέφτω, ε, θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικός ο συντονισμός και χρειάζεται περισσότερος συντονισμός, περισσότερη συζήτηση για αυτό το θέμα. Σε ποιες περιπτώσεις παραδίδουμε όπλα και σε ποιες όχι. Για παράδειγμα η Άννα Γκόμες ανέφερε κάτι πάρα πολύ ε, χρήσιμο. Ένα παράδειγμα που μας δείχνει τις νέες προκλήσεις που έχουν αναδειθεί και πραγματικά ποιο θα πίστευε ότι μια χώρα όπως η Γερμανία που στην ουσία έχει ως αρχή της το ότι δεν παρατηρούμε όπλα σε περιοχές που μαστίζονται από ένοπλες σειράξεις θα εξελιχθεί σε έναν μη κρατικό φορέα. Θα παραδίδει όπλα σε έναν μη κρατικό φορέα όπως τους Κούρδους στο Ιράκ. η οποία είναι μια ομάδα που δεν συγκροτεί όμω κράτο. Πιστεύω λοιπόν πως εν ώψη των εξελίξεων πρέπει και εμείς να επαναθεωρήσουμε τις εφιστάμενες απόψεις μας. Πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα. Επίσης, να σας παραπέμψω στο άρθρο 51 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, το δικαίωμα για συλλογική άμυνα. Απόρρια του οποίου, όπως και ε, βλέπουμε τώρα, είναι αυτό που συμβαίνει. Να λέμε ότι εμείς δεν θέλουμε να λάβουμε μια τέτοια πολιτική απόφαση, να πατήσουμε σε ξένο με τις δικές μας δυνάμεις, Λαμβάνουμε λοιπόν την απόφαση να μην παρέμβουμε, όμως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι ευθύνη όλων μας. Όπως σας είπα, απορρέει από το άρθρο 51. Όλα αυτά είναι μια εξέλιξη η οποία σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Όμως πιστεύω πως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή, όσο δύσκολη και αν είναι, σχετικά με τις εξαγωγές όπλων. Επίσης πιστεύω ότι εκ των υστέρων είναι εύκολο να κρίνουμε. Σίγουρα όμως χρειάζεται να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό όπου θα μπορούμε να κρίνουμε εκ των προτέρων μια κατάσταση και για να γίνει αυτό χρειάζεται ειλικρίνεια. Πρέπει να έρθουμε σε αντιπαράθεση με το εφιστάμενο καθεστώς και να γίνει και μία αξιολόγηση. Φυσικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκομίσουμε συμπεράσματα. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να φανταστώ κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει όπλα στον Ασάντ. Διότι σε σύγκριση με το Ισλαμικό κράτος έχει σκοτώσει 7 φορές περισσότερους εσύρους από ότι το Ισλαμικό κράτος και το κάνει μάλιστα με τρόπο ε, εξίσου βίο και βάναυσο όπως ε, εκείνη και όχι ανοιχτά κιόλα. Γι' αυτό λοιπόν το να στέλνουμε όπλα στον Ασά το θεωρώ απαράδεκτο. Η αιτία φυγής όλων αυτών των ανθρώπων στη Συρία δεν είναι μόνο το Ισλαμικό κράτος. Γι' αυτό πρέπει να ληφθεί, πιστεύω, σοβαρά υπόψη και αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φρόιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το θέμα αυτό. και ειδικότερα όπως το βλέπουμε δεν μορφώνεται στη σημερινή συζήτηση. Θέλω να εστιαστώ σε μία παράγραφο που ανέφερε η Αναγκόμες, αλλά μόνο εν συντομία. Αναφέρομαι στο ζήτημα της διαφάνειας. Λέει εδώ ότι θεωρούμε λυπηρό ότι μόνο 21 κράτη-μέλη υπέβαλαν πλήρη συμμετοχή στην 16η ετήσια έκθεση. Εκφράζεται λύπη του διότι η Ελλάδα δεν παρουσίασε καθόλου στοιχεία, ενώ η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν παρουσίασαν στοιχεία σχετικά με πραγματικέ εξαγωγέ όπλων και η Γαλλία παρουσίασε έναν συνολικό αριθμό για τι εξαγωγέ όπλων χωρί επιμέρου ανάλυση. Πιστεύω ότι ειδικότερα όσον αφορά την Ελλάδα και τη Γερμανία που μέχρι ότου συζητήσαμε το θέμα των προσφύγων και των ρωτών των άσυλο ε, κυριάρχησαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις ζωές μας με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας πιστεύω ότι θα αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία το να μάθουμε τα νούμερα πόσα όπλα έχουν παραδώσει οι Γερμανοί στην Ελλάδα και αν αγόρασε η Ελλάδα τα όπλα αυτά, πόσο τα αγόρασε. Θα πρέπει να σκεφτούμε, να ξέρουμε και το ενδεχόμενο κάποιο είδο κυρώσεων για χώρες που δεν μας παρέχουν τις πληροφορίες ε, τις οποίες ζητάμε, όπως ε, βλέπουμε στην περίπτωση της Ελλάδας. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, I think that ends. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έτσι ολοκληρώνουμε και τη συζήτηση. ως Φροντζουλίτσα και μετά εγώ ίδια βέβαια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλοί λένε, με λένε Φροντζουλίτσα το διαβάζουν σαν να είναι πολωνικό ή κροατικό. Στην πραγματικότητα ονομάζουμε φρουνζουλίκα, όχι φρουνζουλίτσα. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν προσβάλλομαι Είναι, μοιάζουν έτσι κι αλλιώς, δεν είναι και πολύ μακριά το ένα το άλλο. Ήρθα από την Επιτροπή ΝΤΕΒΕ ε, που συνεδριάζει ταυτόχρονα παράλληλα Οπότε προσπαθώ να μοιράσω το χρόνο μου. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκε ότι η Γαλλία δεν θα δώσει τα Μιστράλ στη Ρωσία, τελικά. Όμως κάποιες μεταφορές τεχνογνωσίας, ευαίσθητη τεχνογνωσίας και τεχνολογίες έχει ήδη γίνει από τη Γαλλία προς τη Ρωσία και μην εκπλαγείτε αν δείτε στο μέλλον την Ρωσία να χτίζει, να φτιάχνει συγγνώμη, πλοία που θα μοιάζουν πάρα πολύ στα Μιστράλ. Πρόκειται ένα θέμα το οποίο έρχεται από το παρελθόν αλλά είναι πολύ επίκαιρο και θα παραμείνει στην επικαιρότητα στο μέλλον. Οι εξαγωγές όπλων ε, ενισχύουν την ανασφάλεια σε πολλά μέρη του κόσμου. Γιατί θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα ποιος παραδίδει όπλα και ιδιαίτερα ε, και μεγάλα όπλα στον ε, Ισλαμικό στρατό. Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει. Διότι έχουν πάρει όπλα από τη Συρία, από το Ιράκ, από ορισμένες στρατιωτικές βάσεις αλλά στα χέρια τους φτάνουν τεράστιες ποσότητες ε, ε, πυρομαχικών, αρμάτων, όπλων κλπ. κλπ. Και δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Οπότε είναι φαύλος κύκλος. Καταπολεμούμε πολεμάμε εναντίον του Ισλαμικού στρατού, αλλά υπάρχουν δυνάμεις που το υποστηρίζουν κιόλας, τον υποστηρίζουν κιόλας. Το θέμα του ε, ελέγχου των, εξωτερικών, των εξαγών όπλων θα πρέπει να το βλέπουμε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Ε, δεν υπάρχει πραγματική κέπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να λαμβάνει υπόψη τον έλεγχο των όπλων και τις εξαγωγής όπλων. Υπάρχουν απλώς χώρες που αποφάσισαν να υπογράψουν κάποιες συμφωνίες, άλλες χώρες οι οποίες δεν τις υπέγραψαν, Χώρε χώρες οι οποίες δίδουν στοιχεία, άλλες χώρες οι οποίες δεν δίνουν κανένα απολύτως στοιχείο για τις εξαγωγές όπλων τους κλπ. Στο μέλλον θα έπρεπε λίγο να δούμε ενδεχομένως ε, τις ρίζες των φαινομένων και να εντάξουμε το ζήτημα αυτό στην ΚΕΠΑ. Γιατί οι απειλές και οι προκλήσεις ε, ε, ε, για το μέλλον είναι τεράστιες σε ό,τι αφορά την σταθερότητα και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει οι εξαγωγές όπλων και το εμπόριο όπλων να αποτελέσουν άλλο ένα θέμα διέρεσης, άλλο ένα λόγο διέρεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και μην ξεχνάσουμε και πόσο επηρεάζει και το μεταναστευτικό στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για το ζήτημα αυτό και την έκθεση. Στην έκθεση αναφέρονται οι προκλήσεις. που αντιμετωπίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ανατολική ιτώνια μας. Θα πρέπει οι εξαγωγές όπλων να ειδωθούν και υπό το πρίσμα της εσωτερικής ασφάλειας και υπό το πρίσμα της ασφάλειας των χωρών προς Ανατολάς μας ε, και αυτό θα πρέπει να γίνει στην έκθεση. Ο και είπε ότι είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τις εξαγωγές όπλων στη Ρωσία. Συμφωνώ ότι η επίθεση στην, στη στάδαφος της Γεωργίας ε, ε, ήταν πάρα πολύ σημαντική και θα πρέπει να αξιολογηθεί γιατί ε, έχει περάσει αρκετός χρόνος. Ήδη έχουμε στοιχεία και για την προσάρτηση της Κρυμαίας και θα πρέπει να καταγράψουμε τις παραβιάσεις ε, των ε, κυρώσεων που έχουν επιβληθεί ε, και που είχαμε αποφασίσει από κοινού έναντι της Ρωσίας. Θα πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε σωστά την κατάσταση στην Συρία. Η κατάσταση Συρία αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της ε, προσφυγικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι σημαντικό να δούμε πώς έχουν δράσει οι χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουμε και το τόξο της μετανάστευσης στην υποσαχάρη Αφρική, στο Σάχελ. Εκεί η μετανάστευση γίνεται από οπλισμένες ε, μαφιόζικες οργανώσεις και πολλές φορές και ισλαμικές οργανώσεις <clears throat> που μέσω βίας και με τη χρήση όπλων πιέζουν ε, πρόσωπα και αποκτούν τεράστια κέρδη μέσω αυτού του εμπορίου. Αυτές είναι οι σύγχρονες προκλήσεις και θα πρέπει να τις δούμε στην έκθεση παρόλο ότι ξέρω πως ε, η έκθεση αναφέρεται ήδη σε μέσα από αυτές. Νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση. Ο κ. Γκάλερ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στο σημείο 21. Υπάρχει μια αναφορά λοιπόν στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου εκφράζεται η λύπη για το ότι δεν έχουν δώσει επαρκή δεδομένα. Καταρχάς να σας πω ότι η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων υπόκειται στην εθνική νομοθεσία. Είναι θέμα των εθνικών κοινοβουλίων. Υποθέτω λοιπόν ότι δεν έχουν αποσταλεί ε, επίκαιρα, επικαιροποιημένα δεδομένα, διότι η νομοθεσία στη Γερμανία ή δεν ξέρω μπορεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν προβλέπει κάτι τέτοιο για τις ε, εξαγωγές. Όμως υπάρχει ενδεχομένω μια δυνατότητα εκ των υστέρων σε, όταν πρόκειται για εξαγωγές όπλων από τις προηγούμενες χρονιές να αποσταλούν ε, λοιπόν ε, αυτά τα νούμερα στα Εθνικά Κοινοβούλια. Να σας αναφέρω λοιπόν την άποψή μου. Δεν πιστεύω ότι δεν έχουν αποσταλεί καθόλου δεδομένα, ότι δεν έχουν αποσταλεί επίκαιρα δεδομένα. Στη Γερμανία αυτό είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και τα δεδομένα αυτά είναι απόρριτα. Δεν, ε, ε, δεν ε, ενημερώνονται μάλιστα ούτε τα μέλη του Κοινοβουλίου μας στην Ολομέλεια. Μπορούμε όμως να πάρουμε αυτές τις πληροφορίες για τα προηγούμενα έτη. Εντάξει, ακούγεται πολύ σοβαρό ότι δεν έχουν αποσταλεί καθόλου δεδομένα του χρόνου, θα αποσταλούν όμως. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον ε, κύριο Πιαγλατών για να μας ε, εκφράσει τη δική τοποθέτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εστίασε την προσοχή του σε αυτό το ζήτημα. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναβρίσκομαι μαζί σα μετά από την απρόσθεση τη 14η Ιουλίου που αφορούσε το ίδιο θέμα. Αν μου επιτρέπετε, θα σας ενδιαφέρει φαντάζομαι να σας πω για την αποτελέσματα της πρώτης διάσκεψης ε, που έλαβε χώρα στο Κανκούν του Μεξικό τον περασμένο μήνα. Ε, αφορούσε ακριβώς ε, το ζήτημα που συζητάμε σήμερα αυτή η διάσκεψη ήταν ουσιαστική γιατί οθέτησε της απαραίτητες αποφάσεις ώστε να προχωρήσει το καθεστώς και να εφαρμοστεί η διασκέψη αυτή στην Κανκούν ε, έκανε κάποια διευθέτηση για τη λήψη αποφάσεων, τους οικονομικούς κανόνες και θα επιτρέψει την επαρκή χρηματοδότηση του καθεστώτος και ειδικότερα τις συναντήσεις των κρατών μελών και της γραμματείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το τεράστιο έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί, ειδικότερα από τη γραμματεία. Η διάσκεψη οργανώθηκε από την ίδια τη γραμματεία με επικεφαλή στον Ντενίσα Μιντλαλά από την Ετεφρική για την περίοδο σύσταση της γραμματείας ενός έτους δηλαδή και μετά θα αποφασιστεί ποιος θα είναι ο κανονικός επικεφαλής για τέσσερα χρόνια και η γραμματεία θα έχει έδρα τη Γενέβη. Κάτι σημαντικό όσον αφορά τη διαφάνεια, η διάσκεψη αποφάσισε πρότυπα για τις, υπο... τις εκθέσεις που θα υποβάλλονται. Τα κράτη-μέλα δηλαδή θα πρέπει να συμμορφώνται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις όσον αφορά τις εκθέσεις, ε, συγκεκριμένα πρότυπα, συγκεκριμένες προθεσμίες. Οι εκθέσεις αυτές θα είναι δημοσιοποιημένες. Εμείς αυτό που υποστηρίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δημοσιοποιούνται οι εκθέσει αυτέ αφού γίνεται αλλαγή τη μεταξύ των κρατών μελών, ώστε όλοι στην κοινωνία που ενδιαφέρονται να μπορούν να διαβάσουν αυτέ τι εκθέσει. Οι εργασίε θα συνεχιστούν, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια βάση για τι πρώτε εκθέσει ε, που έχουν προθεσμία το Δεκέμβριο. Καλά λοιπόν είναι τα νέα. Για το μέλλον τώρα η συνθήκη θα δει μεγάλη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δούμε τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα εκεί εστιαζόμαστε. Έχουμε υιοθετήσει τις ε, κατευθυντήριες γραμμές, όπως γνωρίζετε, ώστε να αντικατοπτρίζουν, να αποτυπώνουν και τις κατευθυντήριες γραμμές του ATT, ώστε με ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών να υλοποιούμε τα οκτώ κριτήρια της κοινωνικής θέσης και την εντολή του συνθήκης εμπορίου όπλων. Επίσης ε, έχουμε υιοθετήσει ένα πρόγραμμα σημαντικό με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει αρρωγή σε ορισμένες χώρες εφόσον το ζητήσουν για να ενισχύσουν τα συστήματα ελέγχου εξαγωγής όπλων τους σε συνάρτηση με τη συνθήκη. Κάνουμε λοιπόν πολλή δουλειά επιτόπου στις χώρες αυτές με συγχρηματοδότηση της Γερμανίας και όλες αυτές οι δουλειές που αποσκοπούν στην αποτελεσματική υλοποίηση συνοψίζονται σε μία λέξη που ακούσαμε πολλές φορές σήμερα, διαφάνεια. Διότι ξέρετε πρέπει να είμαστε σαφείς. Προσπαθούμε να είμαστε διαφανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα ε, δεν είμαστε απόλυτα, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αλλά αν δείτε την παγκόσμια εικόνα, η διαφάνεια στις εξαγωγές και εισαγωγές όπλων είναι μάλλον εξαίρεση κανόνας. Διότι σε πολλές άλλες χώρες, εκτός του μπλοκ συγκεκριμένων χωρών, ε, ο εμπόριο όπλων χαρακτηρίζεται από μυστικότητα. Δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία και πολλές χώρες δεν έχουν καμία βούληση, καμία πρόθεση να μοιραστούν στοιχεία. Οπότε αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για την εφαρμογή της συνθήκης. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάμε μερικές ε, χώρες να καταρτήσουν ένα κατάλογο εξαγωγής όπλων το, το βασικό πρώτο βήμα, ε, διαφάνεια, διαφάνεια για ποια ε, εμπορεύματα και πώς ελέγχονται. Όλα αυτά βασίζονται σε ένα κατάλογο ελέγχου στον οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αυτά τα εμπορεύματα. Τι νοείται ως όπλο σε κάθε χώρα. Από εκεί ξεκίνησε η κατάρτιση αυτού του καταλόγου και τους βοηθάμε με αυτό. Και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, η διαφάνεια λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει κόσμο που ενδιαφέρεται να διαβάσει τις εκθέσεις. όταν κάποιος τις ε, εξετάζει, τις ελέγχει, τις αμφισβητεί. Γιατί όπως είπε και η κυρία Γκόμες, έχουμε τις απαιτήσει του νομικού μέσου, τις συνθήκες ας πούμε εμπορίου όπλο, αλλά αν δεν υπάρχει εξέταση, ανάλυση, δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει και κίνητρο για βελτίωση. Και τελικά είναι περιττό το όλο σύστημα, γιατί ξέρετε η διαφάνεια έχει κάποιο ε, επομίζονται κάποιο κόστος για την υποβολή εκθέσεων οι εθνικές αρχές. Το ανέφεραν και πολλοί ευρωβουλευτές ότι η Ελλάδα δεν παρήχε στοιχεία για πέρυσι. Ξέρετε, αυτό μπορεί να είναι και συνέπεια ε, έλλειψης διοικητικών πόρων που έχουμε περικοπεί όταν δεν έχει κανείς πια κόσμο για να συλλέξει τα δεδομένα, να τα συγκεντρώσει και να τα συμπεριλάβει σε μια έκθεση, υπάρχει πρόβλημα, αυτό έχει συνέπεια και οσο αφορά τη διαφάνεια. Όλο αυτό κοστίζει. Δηλαδή πρέπει να επιτευχθεί κάποια ισορροπία μεταξύ του τι μπορούν να αναλάβουν οι εθνικές αρχές και τι έχει νόημα να παραδώσουν ως στοιχεία σε όσους θα εξετάσουν τα δεδομένα. Ε, είναι μια συνεχής διαδικασία αυτή η βελτίωση και επίσης μας ενδιαφέρει να ξέρουμε πού λαμβάνονται οι, οι αποφάσεις για διοδοτήσεις ε, στην Ευρώπη όπως ξέρετε αυτό γίνεται σε εθνικό επίπεδο θα σταματήσω εδώ και ευχαριστώ να απαντήσω τις ερωτήσεις σας. Υπάρχει μια ερώτηση της κυρίας Γκόμες για το τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους δημοσιολαβητές και κατά πόσο ελέγχουμε επαρκώς ε, τα κυνηγητικά όπλα και τα όπλα περαστεχνικά όπλα. Ξέρετε, υπάρχει συνεργασία μεταξύ αστυνομία ε, και τελωνίων με μια προσπάθεια σύγκλησης των πολιτικών ελέγχου των εξαγωγών μεταξύ κρατών μελών. Έχουμε και εμείς μια αρμοδιότητα μερικές φορές αλλά ξέρετε το ζήτημα που έχουμε με τα καλά συνοικοφία παράδειγμα που χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικούς σκοπούς ε, ή για το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το πρόβλημα αυτό έχει περισσότερο να κάνει με τους κανόνες που αφορούν πολίτες ε, όσον αφορά συγκεκριμένα όπλα εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που διαφέρουν μεταξύ κρατών μελών. Δεν έχουν όλα τα κράτη με τους ίδιους κανόνες για το ποια όπλα απαγορεύονται για πολιτικούς σκοπούς. Ε, ε, αυτόματα ή μη αυτόματα σε ορισμένα κράτη απαγορεύονται πλήρω, επίσης είναι και το θέμα των συλλεκτών ε, τα, υπάρχουν οι για τον κατόχων πολυβολών όπλων επίσης έχουμε τα τυφαϊκία τα οποία σε ορισμένα κράτη-μέλη απαγορεύονται εντελώς και σε άλλα επιτρέπονται γιατί οι κανόνες ε, έχουν ακόμα περιθώριο βελτίωσης όλα τα ζητήματα ε, δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες ΚΟΑΡΜ βέβαια και δεν έχουν εξεταστεί ακόμα την ΚΟΑΡΜ αλλά πρέπει να επιληθούν τώρα το κεκτημένο όσον αφορά την κυκλοφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρήση ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα επανεξετάζει το ζήτημα και ελπίζω ε, να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο όσον αφορά το θέμα αυτό. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λατών. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω την εκπρόσωπα από το, την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΣΕΝΤΕ που μου έδωσε το λόγο και τη δυνατότητα να σε ενημερώσω για την εφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την καταπολέμηση τη διακίνηση πυροβόλων όπλων στην Ένωση. Φυσικά, η Γενική Διεύθυνσή μα καλωσορίζει την έκθεση αυτή και την αναφορά στην παράγραφο 6 για την πιθανή αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας που αναφέρατε κι εσείς. είναι η οδηγία 91 σχετικά με την κατοχή από πολίτε πυροβόλων όπλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι, γίνεται αναγκαία αυτή η αναθεώρηση. Όλοι ξέρουμε τι έγινε στο Παρίσι, στην Κοπενχάγη, στη Μασαλία, με τους πυροβολισμούς και όλα αυτά είχαν ένα κοινό, τα πυροβολά όπλα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει θέμα με το ε, κενό που έχουν οι υπηρεσίες πληροφοριών ε, να εντοπίσουν από πού προέρχονται αυτά τα όπλα. Προέρχονται από ληστείες, είναι συνέπεια ε, χρήσης όπλου που βρισκόταν σε αθιστία, επαναχρησιμοποίηση όπλου από πού έρχεται, από τη Μέση Ανατολή, από τη Βόρεια Αφρική. Όλα αυτά είναι μέρος της δουλειά μας στην Γενική Διευθυνσή έτσι ώστε να βελτιώσουμε την εικόνα της κατάστασης. Τώρα σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων πρέπει να σας πω ότι δημοσιεύσαμε μία ανακοίνωση, μία στρατηγική του 2013. Ήταν το πρώτο τέτοιο έγγραφο της Γενικής μας Διεύθυνσης το οποίο αναφερόταν σε πολιτικές δεσμεύσεις και στην πρόσφατη ατζέντα μας για την ασφάλεια. Αναφέρεται το έγγραφο αυτό σε ορισμένες προτεραιότητες. Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καταπολέμηση τη τρομοκρατίας. Εννέα τον αριθμό ήταν αυτέ οι προτεραιότητε Και βασισμένη στι προτεραιότητε αυτέ, η Ευρωπόλ τι χρησιμοποίησε και άρχισε να βελτιώνει την ποιότητα των γνώσεων που έχει. Τώρα υπάρχει ένα σχέδιο δράση που την καταρτήσαμε, το οποίο αφορά στα πυροβόλα όπλα και από νομικής άποψης θα ήθελα να σας ενημερώσω για την ε, τρέχουσα κατάσταση. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι στα τέλη του χρόνου να δημοσιεύσει ένα έγγραφο για την κατοχή πυροβόλων όπλων από πολίτες. Είναι ε, ένα κομμάτι του νομικού πλαισίου λοιπόν της Ένωσης που αφορά την κατοχή, χρήση και μεταφορά όπλων στην επικράτεια της Ένωσης. Η έκθεση η οποία ελπίζω να γίνει δεκτή, να υπερψηφιστεί ως πακέτο, θα έχει στόχο λοιπόν αυτή την ε, αναθεώρηση. Η αναθεώρηση της κατοχής και χρήσης ε, όπλων είναι ένα θέμα που είναι αρκετά επίκαιρο και έχει ε, συζητηθεί ιδιαίτερα της ε, χρήσης επαναδραστηριοποιημένων όπλων. τα οποία μπορούν να επανέλθουν από την αδράνεια με την αλλαγή ενός εξαρτήματος. Με το έγγραφο αυτό επίσης σκοπεύουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια πλήρη αναθεώρηση της ε, κατοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπεύουμε να το πράξουμε αυτό κάποια στιγμή στο 2016, ανάλογα φυσικά και τις εσωτερικές μας ε, διαδικασίες. Τώρα να σας ενημερώσω και για τις διεθνείς μας δραστηριότητες. Καταρχάς με τα Βαλκάνια, η οποία είναι μια περιοχή που ιστορικά έχει χαρακτηριστεί ως πηγή των όπλων αυτών. Έχουμε λοιπόν επαφές με τα Δυτικά Βαλκάνια και έχουμε κάποιες κοινέ επιχειρήσεις που έχουν οργανωθεί. Οργανώθηκε μάλιστα και ένα συνέδριο σχετικά και Επίσης, σκοπεύουμε να έρθουμε σε επαφή με κάποιες χώρες της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται να γίνει η πρώτη συνάντηση την 1η Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να ε, καταρτήσουμε ένα δεύτερο σχέδιο δράσης ε, για την συνεργασία αρχών επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ε, εν λόγω χώρες έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό το πρόβλημα, το κενό που έχουμε σε πληροφορία για το τι γίνεται με τα όπλα. Φυσικά να σας πω κλείνοντας ότι είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βαλέρο. Θέλετε να πάρετε και εσείς το λόγο, να σχολιάσετε τα... τις ανησυχίες, να απαντήσετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις και για όλα τα σχόλια. Ξέρετε. Ελπίζω ότι οι τροπολογίες που θα υποβάλλετε θα συζητηθούν ε, σφαιρικά και θα βρούμε τη λύση. Θα ήθελα να σας διαβάσω από την έκθεση της Europol το, το εξής ε, πυροβόλα όπλα τα οποία προέρχονται από το Μάλι, τη Συρία και τη Λιβύη ήδη κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή μαύρη αγορά και αυτές οι χώρες μπορούν να καταστούν βασικές ε, χώρες προέλευσης παράνομων όπλων. Σελίδα 41 της έκθεσης Europol. Δεν είναι κάτι το οποίο το επινόησαμε εμείς, αναφέρεται στην έκθεση. Δεν αμφισβητώ το γεγονό ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και πολλές χώρες μάλιστα έχουν και τη δική τους αμυντική βιομηχανία. Η πολεμική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε αναπτύχθηκε καταρχήν διότι θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να αμυνθούμε. Αυτό που τίθεται υπό αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια είναι το εξή. Δεν έχουμε πλέον τις ίδιες απειλές στην Ευρώπη με παλιά. Οπότε τα επιχειρήματα για τη διατήρηση της αμυντικής βιομηχανίας είναι πιο πολύ οικονομικά υπό την έννοια ότι δουλεύουν πολλοί άνθρωποι εκεί. Έχουμε πολλές θέσεις εργασίες που παίζονται. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ποιος είναι ο πραγματικός πρωταρχικός στόχος αυτής της βιομηχανίας αυτού του κλάδου. μια, αν πρέπει να διατηρήσουμε την πολεμική βιομηχανία ε, γιατί έχει πολλές θέσεις εργασία και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να τις δώσουμε δικές μας παραγγελίες γιατί δεν έχουμε πλέον τις ανάγκες που είχαμε παλιά ε, αυτή η βιομηχανία θα κινηθεί προς τις εξαγωγές και εκεί χρειαζόμαστε ένα σύστημα ελέγχου των εξαγωγών γιατί υπάρχουν κράτη κράτη, κυβερνήσεις ή ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που έχουν ως καθήκον να διασφαλίσουν ότι δεν πολλούνται όπλα σε χώρες ή φορείς ή οργανώσεις που δεν πρέπει να έχουν όπλα. Εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι αξιόπιστοι αγοραστές. Και νομίζω ότι για αρκετά χρόνια πια δεν κάνουμε την κατάλληλη αξιολόγηση των ενδυνάμει αγοραστών μας. Αυτό είδα εγώ τα χρόνια που δουλεύα στον τομέα των εξαγωγών όπλων. Η βιομηχανία προφανώς θα πουλάει όπλα, αλλά εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτά τα όπλα δεν καταλήγουν σε λάθος χέρια. Κάποιες ερωτήσεις έγιναν για το θέμα των κυνηγητικών όπλων, των ε, όπλων που χρησιμοποιούνται σε αθλητικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις κλπ. Ε, έχουμε επίσης τα ημιαυτόματα όπλα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ελεύθερους σκοπευτές. Θα πρέπει να ε, αυξήσουμε τον έλεγχο σε αυτά τα όπλα. Για τη Σύπρη και τα στοιχεία, τα αρνητικά στοιχεία. Θα έρθω σε επαφή με την Σύπρη ε, και θα ελέγξω τα στοιχεία. Πολύ σύντομα. Άρθρο, το, παράγραφος 21. Ναι, παράγραφος 21. Για το θέμα των πωλήσεων στο εξωτερικό. Καθώς επίσης και για τις ε, ε, πωλήσει ή τι παραδόσει στον Ισλαμικό στρατό. Δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε από παίρνει τα όπλα του Ισλαμικό στρατό. Ε, γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να μπορούμε να ελέγξουμε όλου του κρίκου τη αλυσίδα μέχρι τον τελικό χρήστη. Ό,τι μπορούμε να ελέγξουμε θα πρέπει να το ελέγχουμε. Επίσης τώρα, ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική γειτονία προς τον Νότο και την πολιτική γειτονία προς τον Ανατολά. Ε, μιλάμε για την Αραβική Άνοιξη αναφέρεται ότι δεν είναι, πολύ δεν είναι μόνο αρνητική η αραβική άνοιξη. Εντάξει, σωστά, θα μπορούμε να το διορθώσουμε. Ε, τώρα, ο έλεγχος εξαγωγών κοστίζει. Πράγματι. Και πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να δαπανίσουμε τα ποσά που χρειάζονται έτσι ώστε να πραγματοποιείται πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το κόστος. Ευχαριστώ. Thank you very much. I think we have... Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως έχουμε εξαντλήσει το χρόνο που διαθέτουμε για αυτό το θέμα και θα ήθελα να σας πανθυμίσω άλλη μια φορά την ε, προθεσμία υποβολής τροπολογιών 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν 12 το μεσημέρι. Η δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου και μετά θα ψηφίσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο και να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν, μέλη και προσκεκλημένους. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μποντιλ Βαλέρο, για την προετοιμασία της έκθεσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ανταλλαγή απόψεων με τον Γιάτσε Πιλίτσα, ειδικό απεσταλμένο για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό και θα μας μιλήσει για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάσκεψη του 2015 για την αναθεώρηση της συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων που έλαβε χώρα τον Απρίλιο και το Μάιο φέτος. Έχετε το λόγο. Okay. Now Θα αρχίσουμε λοιπόν τη συζήτηση για το επόμενο σημείο. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρέσβη Μπίλιτσα, κύριο σύμβουλο και ειδικό απεσταλμένο για την ε, μη διάδοση και τον αφοπλισμό. Θέμα είναι η αναθεωρητική διάσκεψη, ένατη αναθεωρητική διάσκεψη για την ε, συνθήκη μη διάδοσης. Έχετε το λόγο κύριε Πρέσβη. Ε, ε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δώσετε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στα πλαίσια της συνθήκης για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων φέτος. Είναι λοιπόν πρέπον το ότι έγινε μια συζήτηση ολομέλεια στις 10 Φεβρουαρίου πριν την ε, διάσκεψη στο Στρασβούργο, όπου είπα ότι εκπρόσωπο Φεντερίκα Μογκερίνη απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό. Και επίσης ε, ήρθε και σε αυτήν την Επιτροπή δύο φορές, στις 29 Ιανουαρίου και τις 16 Απριλίου. Το θέμα αυτό επίσης συζητήθηκε αυτές τις ε, δύο ημερομηνίες. Σίγουρα θα γνωρίζετε ότι παρά τις επίμονες προσπάθειες που καταβάλαμε εδώ και εβδομάδες δεν ήταν δυνατόν να λήξει η διάσκεψη με ένα έγγραφο κοινή συνένεση. Αυτό έγινε εξαιτία των διαφωνιών που υπήρχαν για την ε, ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο η ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν ότι είναι δυνατή μια επίτευξη συμφωνίας για ένα ευρύτερο ε, πλαίσιο θεμάτων ακόμα και με όλες τις διαφορές που έχουν τα επιμέρους κράτη-μέλη δεδομένης της πολυμορφίας της Ένωσης. Τι έγινε λοιπόν στη διάσκεψη. Η ίδια η διάσκεψη έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη τα κεντρικά γραφεία των Ηνωμένων Εθνών μέχρι τις 22 Μαΐου, από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο. Προείδρευσε ο κύριος Φερούκη από την Αλγερία και χορηγός ήταν και 100, από τα 191 κράτη-μέλη ε, συμμετείχαν μόνο ορισμένα 161 από αυτά. Ε, για πρώτη φορά συμμετείχε και το κράτος της Παλαιστίνης το οποίο το 2015 άλλαξε καθεστώς. Επίσης και το Ισραήλ ε, συμμετείχε στη διάσκεψη υποκαθεστώς παρατηρητού. Πρώτη φορά από το 1995. Υπήρχαν αρκετοί διεθνείς οργανισμοί, σε παρατηρητή. η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας από αυτούς. Επίσης όμως και πιο σημαντικά ε, συμμετείχε και η υπηρεσία, ε, η Διεθνής Υπηρεσία Πυρηνικής Ενέργειας ε, από την Βιέννη. Συμμετείχαν λοιπόν οι διεθνείς οργανισμοί με μάλιστα ενεργότατο ρόλο σε αυτή τη διάσκεψη Είχαμε διάφορες ε, παραπλευρές εκδηλώσεις, διαμοιράστηκε υλικό το οποίο είχε σχέση με τον πυλώνα του αφοπλισμού της ε, συνθήκης. Η οργάνωση ε, του, της διάσκεψης είχε ανατεθεί σε τρεις υποεπιτροπές, εκείνη του πυρηνικού αφοπλισμού, εκείνη της μη διάδοσης και της ειρηνικής εφαρμογής της πυρηνικής ενέργειας. Επίσης η διάσκεψη απεφάνθηκε ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν τρία επικουρικά σώματα. Ένα σχετικά με ζητήματα ασφαλεία και άμυνας, ένα με τα, για τα διάφορα περιφερειακά ζητήματα συμπεριλαμβανόμενης της Μέσης Ανατολής και ένα τρίτο επικουρικό σώμα για την, ε, τις ειρηνικές χρήσεις της ατομικής ενέργειας και την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της συνθήκης. Κατά τη διάρκεια των έντονων συζητήσεων αυτές τις τέσσερις εβδομάδες ε, συζητήθηκαν και οι τρεις πυλώνε οι οποίοι συνοψίζονται στο τελικό σχέδιο έκθεσης. Είναι ένα μεγάλο έγγραφο, 184 ε, παράγραφοι βρίσκονται σε αυτό το έγγραφο και ένα επιπλέον μέρος με διατάξεις για περαιτέρω δράση. Όπως ε, ήθιστε με τέτοια έγγραφα που συντάσσονται σε διεθνείς διασκέψεις. Φυσικά δεν είχαν όλα τα συμμετέχοντα κράτη την ε, άποψη ότι συμπεριλήφθηκαν οι δικές τους επιθυμίες. Ιδιαίτερα στο θέμα της εφαρμογής του άρθρου 6 της συνθήκης που σχετίζεται με τον πυρηνικό αφοπλισμό. Εξαιτία ακριβώς των ιδιαιτεροτήτων που προτείνει το σχέδιο για ε, δημιουργία ε, μια ζώνη στη Μέση Ανατολή χωρίς πυρηνικά όπλα ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 169 του τελικού σχεδίου εγγράφου τρία κράτη οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ε, μπόρεσαν να δώσουν τη συνένεσή τους για το τελικό έγγραφο. Έτσι λοιπόν δεν εγκρίθηκε το τελικό έγγραφο. Συγκεκριμένα τώρα για το λόγο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι συμβαλόμενο μέρος στη συνθήκη. Τα 28 κράτη-μέλη είναι συμβαλόμενα μέρη ξεχωριστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθεστώς παρατηρητή, ο οποίος έχει δικαίωμα ε, λόγου. στα συμπεράσματα του Συμβουλίου που εγκρίθηκαν στις 28 Απριλίου 2015 αναφέρονται τα αποτελέσματα και το περιεχόμενο τη ε, διάσκεψη. Σε αυτά τα συμπεράσματα φυσικά δεν συμπεριλήφθηκαν όλα τα στοιχεία, όλε οι εθνικέ θέσει του κάθε ενό από τα 28 κράτη-μέλη. Πολλά από τα οποία μάλιστα έκαναν τις δικές τους ε, δηλώσεις και είχαν ενεργή δράση σε όλο το συνέδριο, σε όλη τη διάσκεψη. Θα ήθελα να σας αναφέρω τώρα εν συντομία την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 Απριλίου, πριν την ε, αρχή λοιπόν της διάσκεψης και θα πάω κατευθείαν στο πώς ενήργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασισμένοι λοιπόν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, πέντε ε, δηλώσεις ανακοινώθηκαν στην διάσκεψη, στη γενική συζήτηση στις 28 Απριλίου, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Φεντερίκα Μογκερίνη, απευθύνθηκε στην Ολομέλεια και στις ε, τρεις κύριες ε, επιτροπές. Υπήρξαν λοιπόν ε, κοινέ δηλώσει σχετικά με τον αφοπλισμό, με περιφερειακά ζητήματα και με την χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Η δήλωση για την Μέση Ανατολή δόθη από τον πρέσβη της Λετωνίας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε δικαίωμα ομιλίας στην περίπτωση αυτή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε τρία εγκεκριμένα έγγραφα εργασία. ένα σχετικά με την πλήρη συνθήκη για τι πυρηνικέ δοκιμέ, ένα άλλο για την πυρηνική ασφάλεια και τι ασφαλιστικέ δικλείδε στη χρήση πυρηνικών. Επίση, διοργανώσαμε δύο ε, εκδηλώσεις, η μία για τη μη διάδοση των ευαλιστικών πυράβλων και μία άλλη για την πυρηνική ασφάλεια. Το τελευταίο, η τελευταία μάλιστα εκδήλωση έγινε με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας. Επίσης παρευρεθήκαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις, κάποιες από αυτές διοργάνωσε η Αίγυπτος και διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πριν το συνέδριο, με τη βοήθεια του Consortium για την μη διάδοση, η Ευρωπαϊκή Ένωση διοργάνωσε ένα σεμινάριο στο Αλγέρι ε, με τη χορηγία του Υπουργείου Εξωτερικών της Αλγερίας και την ε, ενεργό συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργού. Με συμμετοχή των τριών Προέδρων ε, των Επιμέρους Επιτροπών της ε, Διάσκεψης. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο το σεμινάριο και για τον ε, Πρόεδρο της Διάσκεψης αλλά και για όλους τους συμμετέχοντες. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω στο βασικό σημείο που ήθελα να συζητήσουμε σήμερα αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, στην διασκέψη αναθεώρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμφίβολα είναι η πιο πολυπίκυλη από όλε τι ομάδε κρατών που λαμβάνουν το λόγο με συμφωνημένες θέσεις στη διαδικασία. όλε οι άλλε ομάδες κρατών, όπω όπως η P5, το Non-Allied Movement ε, που συμμετέχει ή το NPDI όλοι αποτελούνται είτε από κράτη με πυρηνικά όπλα είτε από κράτη χωρίς πυρηνικά όπλα. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει και τους δύο τύπους κρατών. Τόσο δηλαδή κράτη που είναι ουδέτερα και άλλα που ανήκουν σε κάποια πυρηνική στρατιωτική συμμαχία. Έχουμε κράτη που βασίζονται στην πυρηνική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλα που ε, ε, έχουν επιφυλάξεις για αυτή ή βρισκόνται σε φάση σταδιακής εξάλληψής της. Οπότε είναι μια πολυπίκυλη ομάδα. Και το να, προέρχεται συμφωνημένη, να προέρχονται συμφωνημένες δηλώσεις από μια τέτοια ομάδα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτή τη διάσκεψη. Δώσαμε ένα καλό παράδειγμα επίτευξης δύσκολων συμβιβασμών μεταξύ πολλών διαφορετικών μερών. Ένα παράδειγμα που ακολουθήθηκε σε μεγάλο βαθμό παρότι ένα συγκεκριμένο ζήτημα ε, παρεμπόδισε την τελική συμφωνία. Κυρία Πρόεδρε, η μη επίτευξη συμφωνίας ε, από την Ρευκόν του 2015 σίγουρα δεν είναι κάτι καλό για το παγκόσμιο καθεστώς μη που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά αυτά τα προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να θεωρεί την NPT ακρογωνία λύθη του παγκοσμίου, λίθο του παγκοσμίου και ουσιώδη σημασία για τον αφοπλισμό των πυρηνικών όπλων. Είναι σημαντική για την περαιτέρω ε, ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας για ελληνικούς σκοπούς από τις χώρες εκείνες που θέλουν να ε, αναπτύξουν αυτή την επιλογή. Διατηρούμε λοιπόν τη δέσμευσή μας ε, να διατηρούμε την NPT ως ε, βασικό μέσο για την διασφάλιση της ε, παγκόσμια ειρηνής και σταθερότητας. Επανεβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας και των τριοπυλώνων της ε, συνθήκης και για την τήρηση όλων των σχετικών διεθνών δεσμεύσεων. Ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ε, επιθυμούν οι συντονιστές μας να μιλήσουν κύριε Καλά. Κύριε Ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα έκθεσή σας. Ήμουν και εγώ παρόν στις διαπραγματεύσεις ως μέλος της Γερμανικής και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας και πρέπει να πω ότι απογοητεύτηκα πλήρως. Με απογοητεύσε επίσης η συμπεριφορά ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, ξέρετε τι εννοώ. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο για το μέλλον αυτών των διασκέψεων. Κοιτάξτε τι έγινε στην τελευταία που ως διάσκεψη ήταν μεν πολύ επιτυχής. Ωστόσο πολλά από τα πράγματα που συμφωνήθηκαν εκεί και αποφασίστηκαν δεν υλοποιήθηκαν στη συνέχεια. Η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι τι προοπτικές βλέπετε για το μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, τι θα γίνει στην επόμενη διάσκεψη του 2020. Αναμένεται συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία θα υλοποιηθούν, μάλιστα. Η επόμενη μου ερώτηση είναι η εξή. Τι ρόλο θεωρείτε ότι θα παίξουν οι πολλοί αριθμοί μη κυβερνητικοί οργανισμοί που αναφέρατε ορισμένοι σε κάποιο βαθμό υπήρξαν επιτυχείς. Να σας υπενθυμίσω ε, την υπόσχεση της Αυστρίας. Πώς βλέπετε το μέλλον αυτών των οργανισμών είναι πιο επιτυχής ε, και πιο αποτελεσματική από την επίσημη διάσκεψη. Ε, Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Μαρέκ ωραία, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για δύο ζητήματα της διάσκεψης. Ε, αναφέρθηκε ότι δεν έχουμε συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις μας για την Ουκρανία. σε ό,τι αφορά καταρχήν την συμπερίληψη της Ουκρανίας στο σύνολό της στην συνθήκη. ως ανταπόδοση στην ε, άρνηση διατήρησης πυρηνικών όπλων μετά την πτώση της Σοβιετική Ένωσης. Σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα, θα ήθελα κάποιες περισσότερες εξηγήσεις. Και δεύτερον, κάτι που έχει σχέση με τη μη διάδοση. Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα ως μέσο πολιτικής πίεσης προς τις χώρες που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Αυτό άλλωστε κάνει ε, σε κάποιο βαθμό η Ρωσία που απειλεί χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα ε, ασκεί τέτοιου είδους πολιτική πίεση το έχουμε δει αυτό ε, στο πλαίσιο των τελευταίων διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα στο Μίνσκ θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτό το ζήτημα Πρόεδρος ε, Συμφωνώ και προσυπογράφω αυτή την τελευταία ερώτηση του κύριου Γιούρεκ. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε και για τις συζητήσεις για το πρόγραμμα του Ιράν. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να σας δώσω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ. Α, συγγνώμη κύριος Καν. Ο κύριος Καν έχει το λόγο. Θα είμαι σύντομος. Και εγώ σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε για το κατά πόσον κάνουμε ουσιαστικές ουσιαστική πρόοδο. Οι δικές μου, η δική μου ανησυχία είναι η εξής. Καλωσορίζω τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά πώς θα μπορούσαμε ε, να εξαλείψουμε τα πυρηνικά από τη Μέση Ανατολή ε, γνωρίζοντας ότι μια χώρα τα ε, έχει πυρηνικά όπλα και αυτό οθεί και τις υπόλοιπες να τα αποκτήσουν. Δεύτερον, το θέμα του, του πυρηνικού flashpoint με την Ινδία και το Πακιστάν. Ε, τελευταία έχουν ξαναπαρουσιαστεί εντάσεις στα σύνορα τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση πέραν του να είμαστε παρατηρητές. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Ευχαριστούμε. Δεν είναι το τέλος της συζήτησης όπως φαίνεται. Τσαρστάνο παρακαλώ. Ο κ. Καλά αναφέρθηκε σε μια χώρα που υποθέτω είναι το Ισραήλ η οποία δεν ανεπιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε την κατοχή πυρηνικών όπλων. Να υπενθυμίσω σε όλους όμως ότι το Ισραήλ ουδέποτε υπέγραψε τη συνθήκη, οπότε δεν δεσμεύεται από αυτήν τη συνθήκη τη, της μη διάδοσης και του φοπλισμού. Οπότε δεν λαμβάνει τη βοήθεια που λαμβάνει η Ινδία και το Πακιστάν ως αντάλλαγμα. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά τη συμφωνία με το Ιράν. Είστε ικανοποιημένοι βελτιώθηκαν ε, οι επιβεβαιώσεις, ε, οι απαλληθεύσεις και η παρακολούθηση των τεχνολογιών, ή ε, επιτόπου επιθεωρήσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι το Ιράν θα συμμορφωθεί με τη συμφωνία αυτή, διότι λογικά πρέπει να έχουν γίνει κάποιες σοβαρές βελτιώσεις τώρα, να είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνουν πράγματα μυστικά γιατί, όπως ε, είχε προσπαθήσει το να κάνει στο παρελθόν. Τώρα με τη σύγχρονη τεχνολογία, με τις επιτόπου κάμερες ε, και τον εξοπλισμό μετρήσεων υψηλών επιπέδων ε, ραδιενέργειας δεν υπάρχει πλέον περίπτωση να πειραχτούν από κάποιον ώστε να παραποιηθούν τα στοιχεία που παρέχουν και να είμαστε βέβαια τη σύμφωνοι. Ευχαριστούμε κύριε Βεβίτσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις. Είναι πολύ δύσκολες πρέπει να παραδεχτώ όσον αφορά τις προοπτικές για το μέλλον. Ο κύκλος αναθεώρησης είναι πενταετής. Αυτό σημαίνει ενισχυμένος κύκλος ο οποίος θα θεσπίστηκε όταν επεκτάθηκε, όταν η συνθήκη αυτό ε, και προβλέπονται τρεις προπαρασκευαστικές συναντήσεις ε, για τον κύκλο των πέντε ετών. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι το έτος μετά από τη μεγάλη ε, διάσκεψη αναθεώρησης δεν συμβαίνει τίποτα. Έχουμε δηλαδή ένα έτος απραξίας θα λέγαμε πριν περάσουμε στην πρώτη ρεύκον και στη δεύτερη και στην τρίτη με, μέχρι που φτάσαμε στην ε, διάσκεψη αναθεώρηση του 2015. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι ελπίζουμε ότι το διεθνές περιβάλλον μπορεί να βελτιωθεί από αυτή την άποψη και αναμφίβολα και αυτό περιλαμβάνεται και στην ε, θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χώρες ε, με τα μεγαλύτερα πυρηνικά απλοστάσια όπως η Ρωσική Ομοσπονδία και οι ΗΠΑ, φέρουν ε, ιδιαίτερη ευθύνη στον τομέα αυτών, οπότε σε κάποιο βαθμό είναι συνάρτηση της σχέσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας. Το συνολικό διεθνές περιβάλλον ε, στον τομέα του πυρηνικού αφοπλισμού. Οι πιο πρόσφατες τάσεις φυσικά υπήρξαν απεσιόδοξες για τους λόγους που αναφέρονται και εδώ. οι προτάσεις ε, που τέθηκαν από τον Πρόεδρο Ομπάμα για περαιτέρω διαπραγματεύσεις ε, δεν ε, έγιναν δεκτές από τον Πρόεδρο Πούτιν ούτε από τη Ρωσική Ομοσπονδία γενικότερα. Εμείς επειδή ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα θέλαμε να δούμε πρόοδο στο θέμα αυτό ακολουθούμε την πορεία μας, αλλά, επειδή, αλλά το κατά πόσο θα συμβεί αυτό πριν το 2020, μπορούμε να ελπίζουμε ή να κάνουμε κάτι. Και κάνουμε κάτι όντως, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες για μεγαλύτερη διαφάνεια στον τομέα αυτών. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, διαδραματίζουν σίγουρα κρίσιμο ρόλο. Συνήθως είναι ιδιαίτερα δραστήριες Σημειώσατε ότι ε, συχνά είναι πιο επιτυχής από ορισμένε χώρες, οι ορισμένες διασκέψεις ε, και ρωτήστε γιατί. Κατά την άποψή μου, ορισμένες, οι περισσότερες από αυτές τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις επικεντρώνονται σε ένα ζήτημα μόνο. Γι' αυτό συνήθω ε, είναι πιο εύκολο να σημειώσουν πρόοδο με ένα ζήτημα πιο εύκολο από ότι όταν ασχολείται κάποιο, κάποια κυβέρνηση, ένα διεθνή οργανισμό με ένα πιο περίπλοκο τομέα όπου εξισορροπούνται διάφορα ζητήματα νομικά, πολιτικά και ζητήματα ασφαλεία. Γι' αυτό το λόγο είναι ευκολότερο οι μη κυβερνητικέ οργανώσει να σημειώσουν κάποια πρόοδο από τι διασκέψει τη εκδηλώσει από ότι τα κράτη-μέλη αλλά ας μην απελπιζόμαστε. Είναι εμπόδιο όπως ανέφερα, αλλά η συνθήκη επιβίωσε παρόμοιων ε, προβλημάτων και στο παρελθόν. Εγώ εκ μέρους της χώρας μου συμμετείχα στην ε, διάσκεψη αναθεώρηση του 2005 που ήταν πολύ χειρότερη από, κατά δική μου αξιολόγηση από τη φετινή. Και η συνθήκη και το καθεστώς ε, έχουν επιβιώσει όλων αυτών των προκλήσεων και το 2010 καταφέραμε να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα και πολλά αποτελέσματα όπως τονίσατε ήταν πολύ καλή διάσκεψη και υπερβολικά καλή γιατί θα είναι δύσκολο να τα υλοποιήσουμε όλα εντός πέντε ε, και ενώ οι νομικοί μπορεί να αμφισβητήσουν σε ποιο βαθμό ορισμένε υποχρεώσεις παραμένουν σε ισχύ ή όχι αποτελούν κομμάτι ενός κεκτημένου μη διάδοσης Οπότε δεν πιστεύω ότι ήταν μάταια όλα. Πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη οπτική. Η Ουκρανία είναι ένα από αυτά τα μελανά σημεία του σημερινού κόσμου όσον αφορά την ασφαλεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και εγώ είχα το προνόμιο να εκφωνήσω αυτή τη δήλωση στην πρώτη κυρία Επιτροπή της διάσκεψης που ασχολήθηκε με τον αφοπλισμό. Φυσικά η Ουκρανία ε, ξέφρασε μια ισχυρή άποψη. Το ίδιο και άλλες χώρες ε, ε, αναφερόμενοι στο γεγονός ότι το μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994 το οποίο σχετίζεται με το γεγονός ότι αποφάσισε να γίνει μέλος του NPT η Ουκρανία ως κράτος χωρίς πυρηνικά όπλα έχει παραβιαστεί. Ήταν πολιτική βέβαια η δέσμευση αναμφίβολα και όχι νομική και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ιδιαίτερα σαφής σε αυτό και υπήρξε ιδιαίτερα σαφής εννοώ για το θέμα της Κρυμαίας αλλά και για το θέμα των, ε, της υποχρέωσης του διεθνούς δικαίου και των υποχρεώσεων στον τομέα αυτό της μη διάδοσης και του αφοπλισμού. Το ζήτημα των ε, στρατιωτικών δογμάτων που συζητήσατε, που αναφέρατε, ναι, συζητήθηκε, αλλά από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ορισμένοι επέκριναν εθνικά δόγματα, άλλοι ανέφεραν συμμαχικά δόγματα όπως το ΝΑΤΟ και το πυρηνικό δόγμα φυσικά συζητήθηκε από ορισμένου. Ο ρόλος που έχει διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίλυση για το, όσον αφορά το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα αναγνωρίστηκε στη διάρκεια αυτής της διάσκεψης και θα έλεγα ότι βελτίωσε το περιβάλλον των συζητήσεων παρότι έγινε πριν από την συνολική ε, την τελική ε, συμφωνία ε, ήταν όταν είχε πραγματοποιηθεί η ενδιάμεση συμφωνία οπότε έλαβε πολύ θετικά σχόλια από τα κράτη-μέλη που συμμετείχαν στη διασκέψη και έλαβε πολλά εύσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και για το ρόλο που διαδραμάτισε η ίδια μαζί με την υπατή εκπρόσωπο στην επίλυση του ζητήματος αυτού. Τώρα θα περάσω στο ερώτημα για την επαλήθευση τη στήριξη αυτής της σύμβασης, αλλά δυστυχώς ε, δεν μπορώ εγώ να σας ε, διασφαλίσω ότι ακολουθούνται οι μέθοδοι επαλήθευση. Ε, αυτό είναι δουλειά του Οργανισμού ατομική ενέργεια στην Βιέννη και πιστεύω σήμερα ότι ο απεσταλμένο Γιουκέ Αμάνο κάνει αναφορά στα κράτη-μέλη για τα αποτελέσματα τη επισκεψή του το Σαββατοκυριακό στο Ιράν αλλά προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει το κεντρικό ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού ε, Ατομικής Ενέργειας και έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητες που έχει. Παρέχουμε και τεχνολογίες και ε, χρηματοδότηση στην ΑΕΕ σε ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως πυρηνική ασφάλεια αλλά και ασφαλιστικές δικλείδες και επαλήθευση. Είναι από τους βασικούς ε, χρηματοδότες ε, του οργανισμού η Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε είναι ρόλος και του οργανισμού να καθισκάζει τη διεθνή κοινότητα ότι πραγματι υλοποιείται ορθώς αυτή η συμφωνία όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του ΙΡΕΝ. Τώρα για τη Μέση Ανατολή η ζώνη χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής ε, όπως ανέφερα Παρότι είμαστε ακόμα στο σχέδιο εγγράφου, αυτό το κομμάτι του εγγράφου είναι πολύ σημαντικό. Παρότι έχει βέβαια υιοθετηθεί επίσημα. Το ζήτημα αφορούσε κυρίως ε, τη διαδικασία και όχι το τελικό αποτέλεσμα. Διότι το γεγονό ότι εμείς θέλουμε η περιοχή αυτή να απαλλαχθεί από όλα τα όπλα μαζικής καταστροφής είναι κλασική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με την οποία συμφωνούν και πολλοί άλλοι. Αυτός είναι ο γενικότερος στόχος. Το ζήτημα όμως είναι πώς ε, τέτοιες περιοχές ε, αρχίζουν να υπάρχουν. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένες τελευταίες γραμμές από την Επιτροπή Αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών που επισημαίνει ότι η ζώνη αυτή πρέπει να βρίσκει σύμφωνε όλε τι χώρε ε, τη περιοχή και όχι να επιβάλλεται από, από άλλε χώρε. Να είναι εθελοντική ε, κίνηση όλων των χωρών τη ε, περιοχή. Και εκεί έγινε το πρόβλημα με τι συγκεκριμένε διαδικασίε που αποφασίστηκαν, που προτάθηκαν στο σχέδιο γράφου προ απόφαση. Πώ δηλαδή μια διάσκεψη για το θέμα αυτό θα μπορούσε να συγκληθεί και από ποιον. Όσον αφορά την ιδιότητα μέλους του Ισραήλ, αλλά και της Ινδίας και του Πακιστάν ε, στην συνθήκη μη διάδοσης είναι σίγουρα κάτι που υποστηρίζουμε την ε, παγκοσμιοποίηση αυτή της συνθήκης και για άλλα καθεστώτα όπως τη συνθήκη των χημικών όπλων αλλά και για τη συνθήκη φυσικά της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων συμπεριλήφθηκε μια ρήτρα στο, σχέδιο του τελικό, στο τελικό σχέδιο του γράφου και είναι όπως είπα και κομμάτι τη ε, ευρωπαϊκής θέσης. Εμείς διεξάγουμε διάλογο με όλες αυτές τις χώρες για τη μη διάδοση, τον αφοπλισμό, τα ζητήματα πυρηνικής ασφάλειας και τους προσφέρουμε επίσης και αρρωγή από ε, τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλλά και μέσω της κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Το Ισραήλ λοιπόν, ε, το Πακιστάν και η είναι μόνιμοι συνομιλητέ μα σε αυτά τα πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Κύριο έχει το λόγο. Πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος η Ρωσία να εγκαταλείψει τη συνθήκη. Χαζή ερώτηση είμαι αλλά Σε Αυτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω το θέμα της Ρωσίας σε σχέση με τον ΝΑΤΟ και τα σχετικά έγγραφα. καταρχάς ε, αποτελεί κατάφορη παραβίαση της αξιοπιστίας και είναι μια ένδειξη της αποτυχίας της ε, ένατης αναθεωρητικής διάσκεψης αυτό ότι δηλαδή οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί στην Ουκρανία μετά από το μνημόνιο της Βουδαπέστης ε, δεν τηρήθηκαν και ανταυτόν μάλιστα δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το δόγμα πολέμου που συμπεριλαμβάνει και πυρηνικές επιθέσεις. Το λεγόμενο ρωσικό δόγμα. Και αυτό έγινε μετά την υιοθέτηση αυτού του δόγματος και ακολούθησε φυσικά η προσάρτηση εδαφών. και εδαφών της Γεωργίας και φυσικά η προσάρτηση της Κρυμαίας υπό την απειλή πολέμου εναντί άλλων χωρών. Με άλλα λόγια λοιπόν η Ρωσία προσέβαλε το δικαίωμα αυτοδιάθεσης κυρίαρχου κράτους. ενώ ένας από τους όρους ε, προσάρτησης, ε, εισχώρησης μάλλον στο ΝΑΤΟ είναι η ελεύθερη βούληση των κυριαρχών κρατών. Υπάρχουν προβλήματα λοιπόν και αυτό κάνει τη διαφορά. Παρακαλώ, απαντήστε. Σχετικά με το ρωσικό στρατιωτικό δόγμα. Να πω ότι σίγουρα δίχως αμφιβολία έχει εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις πολλά χρόνια. Έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει βέβαια το ρωσικό δόγμα τα τελευταία χρόνια και μαζί με αυτό και, το, και τα όρια χρήσης τους. Έχει αλλάξει λοιπόν και το σύστημα συναγερμού και ενεργοποίηση πυρηνικών όπλων σε περιπτώσεις ε, έκτακτη ανάγκης, για παράδειγμα Ουκρανία και την προσάρτηση της ε, Κρυμαία. Αυτό ίσως θα το παρατηρήσατε και με τις ενέργειε των ε, διπλωματών που συμμετείχαν στο, στη διάσκεψη. Τώρα σχετικά με το αν υπάρχει κίνδυνο να αποχωρήσει η Ρωσία από τη συνθήκη μη διάδοση. είναι πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς ε, το μέλλον δεδομένων των ε, συνθήκων και όλων των εμποδίων. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω κάποιον τέτοιο κίνδυνο στο άμεσο μέλλον. Η Ρωσία είναι ένας ε, πολύ σημαντικός παίκτη, είναι ένα κράτος που διαθέτει πυρηνικά και συμμετέχει σε αυτήν την συνθήκη. Πρέπει να μας ανησυχούν άλλες συνθήκες, ιδιαίτερα η ενδιάμεση συνθήκη για τις πυρηνικές δυνάμεις, η συνθήκη INF χάρη στην οποία η Ευρώπη κατέστρεψε πάνω από 3.000 πυρηνικές κεφαλές ή πυράβλους με βεληνικές από 500 έως 5.000 χιλιόμετρα, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν οπλισμένοι με πυρηνικές κεφαλές. Η διάδοση λοιπόν αυτών των πυράβλων είναι ένα πρόβλημα εκτός ε, των ανταφών της Ευρώπης είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει έλλειψη νομικών δυνατοτήτων, υπάρχουν κάποια μέσα που υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κώδικας της Χάγης για παράδειγμα, ε, τον οποίο στηρίζουμε και εμείς. Υπάρχουν, υπάρχει διπλωματική οδός, όμως ε, τα μέτρα αυτά είναι περισσότερο μέτρα διαφάνειας ε, παρά μια συνθήκη δεσμευτική. Επίσης, ε, μην ξεχνάμε και το καθεστώ ελέγχου, μέσω του οποίου ορισμένε χώρε προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωση τη της ε, τεχνολογίας πυράβλων που μπορεί να δράσει αποσταθεροποιητικά. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη λοιπόν για την Ευρώπη και υπάρχουν ε, σίγουρα κάποιες κατηγορίες οι οποίες, τις οποίες εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ προς τη Ρωσία και το αντίστροφο και εμείς σίγουρα προσπαθούμε να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη να ε, συζητήσουν. Η συνθήκη αυτή υπεγράφει όταν η Ρωσία ήταν ακόμα Σοβιετική Ένωση και τώρα υπάρχουν άλλα κράτη που έχουν διαδεχθεί λοιπόν τη Σοβιετική Ένωση, Λευκορωσία κτλ. Αυτά λοιπόν για την ανησυχία σας σχετικά με την αποχώρηση από το συνθήκη μη διάδοση. Ε, μην ξεχνάμε τις άλλες εξίσου σημαντικές συνθήκες, όπως την ενδιάμεση συνθήκη. Είναι εξίσου σημαντικές για την ασφάλεια και τον αφοπλισμό των πυρηνικών κρατών. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Ίσως ο κύριος Φρόιντ θα ήθελε το λόγο. Όχι. Κύριε Στετίνα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση. Μπορώ? Κύριε Πρέσβη, έχετε κάποια στοιχεία σχετικά με τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Για παράδειγμα, για νάρκες, με τη χρήση λοιπόν τέτοιων όπλων από τρομοκράτες με την κατάχρηση καλύτερα τέτοιων όπλων. Thank you. Uh, Μπορείτε να μας διευκρινίσετε λίγο την ερώτησή σας. Κύριε Στατίνα, μιλάτε για χρήση τακτικών όπλων ή ε, Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω τον πρεσβή αν έχει πληροφορίες για το γεγονός ότι πυρηνικά τακτικά όπλα όπως ατομικές νάρκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες, αν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. translation was misused by by terror. Misused it is the right expression. Uh, ambassador. Ναι. Ο κύριος Πρέσβης. Δεν έχω τέτοιου είδους στοιχεία ή πληροφορίες για κατοχή, περικατοχής ή σχεδίων χρήσης ε, τακτικών πυρηνικών όπλων από τρομοκρατικές ομάδες. τέτοια όπλα ονομάζονται υποστρατηγικά πολλές φορές, υποστρατηγικά πυρηνικά όπλα. Ε, καλό να το έχουμε στο μυαλό μας. Κάποιοι, κάποιοι αμφισβητούν και την ύπαρξη τέτοιων ε, όπλων. Η, ε, η οποιαδήποτε πυρηνική έκρηξη θα έχει στρατηγικό χαρακτήρα έτσι κι αλλιώς ε. στο παρελθόν Είχαμε χιλιάδες έως και δεκάδες χιλιάδες ε, τακτικά πυρηνικά όπλα ε, όπως ε, όλμους, βόμβες ελεύθερης πτώσης, ορολογιακές βόμβες κλπ. στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά χάρη στο τέλος του ψυχρού πολέμου η ύπαρξή τους περιορίστηκε πολύ μάλιστα υπογραφικές και συμφωνίες και διμερείς ε, ε, ε, διακανονισμοί μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας και κάτι που δείχνει τη μείωσή τους. τώρα, λίγα πράγματα, για σε λίγα πράγματα μπορούμε να συμφωνήσουν όλοι. Ένα από αυτά είναι η PNI, Presidential Nuclear Initiatives, δηλαδή οι πυρηνικές προεδρικές ε, πρωτοβουλίες, δηλαδή μια σειρά μονομερών ε, αλλά συντονισμένων δηλώσεων από πλευράς ε, Πρόεδρου των ΗΠΑ και Πρόεδρου της Ρωσίας, έτσι ώστε να αποσυρθούν τέτοιου είδους όπλα σε κάποιες κεντρικές αποθήκες. Με άλλα λόγια, ότι δεν θα βρίσκονται σε στρατιωτικές μονάδες που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, αλλά σε κάποια κεντρικά υπόστεγα, αποθήκες κλπ. Σε θέσεις που είναι καλά φυλασσόμενες έτσι ώστε να μην πέσουν στα χέρια τρομοκρατών. Αυτές οι πρωτοβουλίες, οι PNIs, ε, είναι πρόσδεκτες και ελπίζουμε ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται συμπεριλαμβανομένες και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Δύο... Α, πολλοί μπορούν να πούν ότι δεδομένου ότι ήταν συντονισμένες, ε, ότι αυτές οι συντονισμένες προεδρικές μονομερείς δηλώσεις ισοδυναμούν με μια διεθνή συμφωνία. Τώρα, όλα τα πυρηνικά όπλα ε, θεωρούνται ένα και το αυτό από τη συνθήκη μη διάδοσης, ε, αλλά για μας εδώ στην Ευρώπη έχετε δίκιο, τα τακτικά πυρηνικά όπλα, που είναι πολύ λίγα στην ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ευτυχώς, περισσότερα, πολύ περισσότερα στην, στο ευρωπαϊκό κομμάτι της Ρωσικής Ομοσπονδίας χωρίς να ξέρουμε πώς ακριβώς. Αυτό λέω είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας. Μια απειλή και ένα κίνδυνο τον οποίο θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Προσπαθούσα να καταλάβω αν πρόκειται για κατοχή ή ε, χρήση ή ε, κατάχρηση. Είναι ο εξής. Ε, αν χρησιμοποιείται οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο, ε, θα, η χρήση αυτή θα εντοπιστεί αμέσως από τους ε, δορυφόρους και τον εξοπλισμό που παρακολουθεί. Οπότε είτε είσαι τρομοκράτης είτε είσαι κράτος δεν μπορείς κρυφά να προκαλέσει έκρηξη τέτοιου όπλου. Δεν έχω δίκιο. γιατί ε, θα ήταν ε, πολύ ανησυχητικό κάποιο να μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο όπλο χωρίς να το μάθει όλος ο κόσμος. Ε, μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε. all... Καταρχήν να κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε ένα πυρηνικό όπλο και σε μια εκρηκτική ε, διάταξη από αυτές που ονομάζουμε dirty bombs, βρώμικες βόμβες θα ήταν ε, μια τέτοιου είδου διάταξη έχει ένα σύνηθες γρηκτικό ε, υλικό εμπλουτισμένο με κάποιο πυρηνικό υλικό. Ε, αυτό είναι κάτι πολύ χαμηλότερο σε επίπεδο από ένα πραγματικό αυθεντικό πυρηνικό όπλο, έτσι προφανώς. Ε, έχετε δίκιο ότι η τεχνολογία επιτρέπει την άμεση, τον άμεσο εντοπισμό, την άμεση ανείχνευση πυρηνικών εκρήξεων και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και ένα, με χρηματοδότηση ένα σύστημα που είναι το Διεθνές Σύστημα Παρακολούθησης του, της εφαρμογής της συνθήκης απαγόρευσης πυρηνικών δοκιμών που έχει τη γραμματεία της, της στη Βιέννη. Η ίδια η συνθήκη δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Το 2016 θα γιορτάσουμε την 20η επέτειο του ανοίγματος συμφωνίας σε υπογραφή. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν ε, επικυρώσει. Ε, υπογράψει και επικυρώσει, απαγορεύει τις πυρηνικές δοκιμές και τις πυρηνικές ε, κρίξεις, όμως ε, ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε η συνθήκη δυσκολεύει πολύ την έναρξη εφαρμογή της, διότι απαιτεί την επικύρωση της και από τις 44 χώρες που καταγράφονταν στο παράρτημα. Τότε που διαπραγματευθήκαμε αυτή τη συνθήκη ήταν οι χώρες οι οποίες εν δυνάμει θα μπορούσαν να ε, έχουν πυρηνικά όπλα. Οκτώ δεν την έχουν υπογράψει. Νομές Πολιτείες, Κίνα ε, δεν την έχουν επικυρώσει μάλλον παρόλο που την υπέγραψαν. Το Ιράν επίσης, το Ισραήλ. Χώρες οι οποίες δεν έχουν, δεν καν ε, μέρη της ε, συνθήκης μη διάδοσης. Οπότε ε, δεν είναι εύκολο να μπει σε λειτουργία. Όμως η συνθήκη αυτή προβλέπει ένα σύστημα παρακολούθησης, επιτήρησης, το οποίο υπάρχει. Έχει δημιουργηθεί, είναι πολύ προηγμένο τεχνολογικά και έχει σεισμογραφικούς ε, καταγραφικούς σταθμούς ε, αλλά και ε, άλλους τύπου υπόγειους, συγγνώμη, υδρα, ε, συ, ε, σταθμούς ε, κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και, ε, και εντοπίζει μικρές εκρήξεις, μέχρι και μικρές εκρήξεις, αλλά όχι μόνο πυρηνικές. Για παράδειγμα, ανείχνευσε τις εκρήξεις στο υποβρύχιο, ρωσικό υποβρύχιο Κούρσκ, παρόλο που δεν είναι πρόκειτο για πυρηνικές ε, εκρήξεις. Το υδροακουστικό σύστημα ήταν τόσο ευαίσθητο που εντόπισε, ανείχνευσε και τις δύο εκρήξεις του υποβρυχίου Κούρσκ. Επίσης, ε, πυρηνικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας έχουν εντοπιστεί και έχουν αξιολογηθεί από αυτό το σύστημα. Οπότε για να σας απαντήσω ναι, πιστεύω ότι είναι σχεδόν αδύνατον να χρησιμοποιήσει κανείς ένα πυρηνικό όπλο ακόμα και μικρής απόδοσης ε, χωρίς να εντοπιστεί, χωρίς να ανοιχνευθεί, ακόμα και αν κάτι τέτοιο συμβεί στη Σαχάρα ή οπουδήποτε άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη για αυτήν την ε, πληρέστατη απάντηση στα πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που σας ετέθησαν. Νομίζω πως εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτό το σημείο της της διάταξης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή συνεδρίαση και σας παρακαλώ αύριο το πρωί να είστε και πάλι εδώ στις 9. Ευχαριστώ πολύ.